Uh, very um, Καλημερίζω όλους. Ξεκινάμε με το δεύτερο τμήμα της συνεδριάσεώς μας για αυτό το μήνα. Έχουμε αρκετέ σημαντικές ψηφοφορίε στι 9 και 45, αλλά πριν θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για μια έκθεση πολιτικής πρωτοβουλίας για την προστασία των καταναλωτών και της υπηρεσίας κοινή ωφέλεια. Θα καλωσορίσω τον κύριο Βίντεν είναι η πρώτη του έκθεση σε μας. Βλέπω ότι έχω και την κυρία Γκάλ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η κυρία Γκέπχαρτ και εγώ που είμαι πολύ συχνά ε, σκιώδης για την ομάδα μου και βέβαια από τους φιλελευθέρους δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή, ίσως έρθουν αργότερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, πριν το κάνουμε αυτό, να καλωσορίσω και τους ακροατές μας ή θεατές μας ε, στο διαδίκτυο και σας θυμίζω ότι υπάρχει ένα καινούριο περιοδικό της Επιτροπής μας, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε διαδικτυακά. Θα καλέσω λοιπόν τον κύριο Βίντεν να παρουσιάσει την έκθεσή του και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Θα πάρουν το λόγο πρώτα οι σκιώδεις. Να καλωσορίσω επίσης και δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεσή σας, κύριε Βίντεν Χόλτζερ. Έχουμε την κυρία Μπλουμ από την Γενική Διεύθυνση Σάνκο που έρχεται πολύ συχνά. και τον κύριο Ποτσμάρσκι από την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο αργότερα να μπορέσετε να σχολιάσετε την έκθεση. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό νομίζω αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και μια βασική συζήτηση η οποία ενδεχομένως να έχει και πολιτικό χρώμα. Θα ήθελα καταρχάς να αναφέρω τέσσερα σημεία σε ό,τι αφορά το αιτιολογικό. Νομίζω ότι καταρχάς έχουμε διάφορες, ε, διάφορους ορισμούς. Ο όρος Φορέα υπηρεσιών κοινή ωφελία δεν έχει οριστεί σε επίπεδο ένωση και χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και στα κράτη-μέλη άλλωστε. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια σύγχυση σε ό,τι αφορά τον ορισμό του όρου. Και αναρωτιέται λοιπόν κανείς κατά πόσον θα χρειαζόμασταν καν μια οδηγία. Αφετέρου υπάρχουν και πάρα πολλά κοινά σημεία τα οποία είναι θεμελιωδούς σε σημασία για την κοινωνία και τη ζωή του ανθρώπου. Είναι λοιπόν θέματα τα οποία πλήττουν και αφορούν τους καταναλωτές. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να διαλευκάνουμε το τοπίο σε ό,τι αφορά τον ορισμό του όρου. Είναι επίσης μια πολύ πολιτική συζήτηση αυτή, η οποία συνεχίζεται τα τελευταία 15 χρόνια. Κατά πόσον τα θέματα των μέτρων απελευθέρωσης έχουν θετικές επιπτώσεις. Διαπιστώνω ότι τα αποτελέσματα της ελευθέρωσης δεν ήταν αμυγός θετικά. Δεν ήταν αμυγός υπέρ του συμφέροντος των καταναλωτών. Άρα και από την ε, οπτική αυτή γωνία σημαντικό είναι να αναλογιστούμε με προσοχή προς τα που θέλουμε να εξελιχθούμε. Αυτό που για μένα είναι καθοριστικό ερώτημα είναι οι καταναλωτές. Και νομίζω ότι έχει νόημα αυτή η πολιτική συζήτηση να περιοριστεί σε πρώτη φάση σε ό,τι αφορά θέματα του καταναλωτή. Να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τα πιο βασικά στοιχεία και γι' αυτό λοιπόν επικεντρώθηκα σε τέσσερις μεγάλους τομείς. Γιατί εδώ θεωρώ ότι έγινε τα πιο βασικά καθοριστικά σημεία. Να υποδείξω και ένα τέταρτο θέμα. Προφανές, αρκετά. Σε καιρούς κρίσης, όπως αυτούς που διανύουμε σήμερα, υπάρχει πάντα μια συζήτηση για το κατά πόσο χρειάζεται μεγαλύτερη ρύθμιση, κατά πόσο χρειάζεται κάποια βελτίωση των πολιτικών και αντιμετωπίζουμε και χρηματοοικονομική πίεση από, από ό,τι γνωρίζετε. Ακριβώς λοιπόν επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το θέμα της καθολικής ε, φροντίδας μέσω των ε, υπηρεσιών κοινή ωφέλεια να μην εγγυάται. Αυτό θα διασφαλίσει και την κοινωνική συμπερίληψη. Ανέπτυξα λοιπόν κάποιες γενικές αρχές, κάποιες γενικές αξιώσεις, οι οποίες στο σκοπό έχουν να διασφαλίσουν θεμελιώδη και να εναρμονίσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεμελιώδη δικαιώματα του καταναλωτή σε ό,τι αφορά αυτές τις υπηρεσίε κοινή ωφέλεια. Η συζήτηση που διεξάγεται συνεχώς για ένα κοινό πλαίσιο υπηρεσιών λύσεων ωφελία. ασφαλώς και περιλαμβάνει διάφορα αμφιλεγόμενα και ακαθόδη θέματα, μια και είναι και θέμα επικουρικότητας σε μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει και μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τι ε, Ευρωπαϊκές ενώσει σημαντικό είναι να συμμετάσχουν και οι οργανώσεις ε, των καταναλωτών, οι κοινωνικές ε, ομάδες. Και επίσης ε, πολύ σημαντικό είναι μαζί με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να τονίσουμε και να ορίσουμε μέσα στον τρόπο τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και να προβλεφθούν ειδικέ ρυθμίσεις. Τώρα, στο θέμα της ενέργειας. Εδώ διαπιστώνουμε ότι με τις τρέχουσες εξελίξεις δεν ισχύουν αυτά που ίσχυαν αυτά που επιθυμούσαμε πριν από 10-15 χρόνια. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η ενεργειακή ένδυα. Θα ήθελα να το θέσω ιδιαίτερα αυτό. Δεν είναι ουδέτερη μόνο η ενέργεια. Το θέμα που τίθεται είναι και η βιωσιμότητα της ενέργειας. Επίσης αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι για τους καταναλωτές είναι όλο και πιο δύσκολο να συγκρίνουν τις ε, τιμές της ενέργειας στην αγορά όπως διαμορφώνεται. Υπάρχει μια συμμετρία σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Το οποίο φυσικά δεν ωφελεί την αγορά. Έχει να κάνει και με τα δικαιώματα πληροφόρησης ε, των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχει μια επισκόπηση σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες αυτές και σε ό,τι αφορά την πραγματικό ύψος των τιμών της ενέργειας. Όλα αυτά από κοινού θα πρέπει λοιπόν να συζητηθούν. Για τις τηλεπικοινωνίες. Το θέμα είναι να είναι ανοιχτό και ουδέτερο το διαδίκτυο σε ό,τι αφορά και την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών που είναι ιδιαίτερη σημασία. Η κινητικότητα των δεδομένων επίσης. Η δυνατότητα μεταφοράς τους. Σε ό,τι αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, το βασικό θέμα είναι η ε, καθολική κάλυψη και της υπαίθρου που συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα και σε ό,τι αφορά τις εργασιακές συνθήκες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές σε ό,τι αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, τώρα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ενίσχυση των δικαιωμάτων των ε, καταναλωτών, αλλά όχι σε ό,τι αφορά τις κοντινές αποστάσεις συγκοινωνίας. Και εδώ λοιπόν είναι σημαντικό το θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα των ε, δημόσιων συγκοινωνιών για μικρές αποστάσεις. Και σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη και τον δημοκρατικό παράγοντα, δημογραφικό παράγοντα. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Να μην αποκλείονται κάποιοι πολίτες από τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτά λοιπόν εν συντομία σε ό,τι αφορά την έκθεση που έχετε ενώπιόν σας. Προσβλέπω και στις μελλοντικέ συζητήσεις, οι οποίες και ελπίζω να είναι αμφιλεγόμενες και να οδηγήσουν σε παραγωγικά αποτελέσματα, επικοδομητικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Good. Well, thank you very much indeed. Now. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι θα ακολουθήσει η συζήτηση ήδη να σας ευχαριστήσουμε για το έργο σας. Το ζήτημα με τις ε, <clears throat> γνωμοδοτήσεις ίδια πρωτοβουλία είναι πάντα το περιορισμό στην έκταση τους, αλλά νομίζω καταφέρατε να αξιοποιήσετε το διαθέσιμο χώρο. Κύριε Καλπέλτ, έχετε πρώτα το λόγο, μέρος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με ικανοποίησε η προσέγγιση του συναδέλφου που ήταν ιδιαίτερα αναλυτική. Θεωρώ το θέμα σημαντικό και η πρότασή σας μπορεί να είναι χρήσιμη όχι μόνο για τις οργανώσεις των καταναλωτών, αλλά επίσης για τους πολίτες, για τα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις. Ο εισηγητής έχει καταγράψει τις προτεραιότητες, την ενέργεια, τις, δημόσιες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. οι πολίτες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, όπως ε, και αυτό ε, ε, οδηγεί σε μεγαλύτερη ανάγκη για διαφάνεια και τη δυνατότητα σύγκρισης των πληροφοριών. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με τον εισηγητή στα εξή σημεία. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την μεγαλύτερη δυνατή προστασία του καταναλωτή, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, οργανώσεις προστασίας του κανατολωτή ισχυρές και λειτουργικές. Θα πρέπει να υπάρξει ένας ορισμός των οργανισμών κοινή ωφέλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και η παροχή δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Πρώτα απ' όλα, για το ζήτημα της ενέργειας. Συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή όσον αφορά τον τομέα το, ζήτημα της απελευθέρωσης του τομέα αυτό. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, κυρίως όσον αφορά την τιμολόγηση και την μετακύληση του κόστους προς τους καταναλωτές, γιατί δημιουργούνται μονοπόλια σε αυτό το τομέα και αυτό προφανώς υπονοβεύει τα δικαιώματα του καταναλωτή. Υποστηρίζω επίσης την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που είναι πιο βιώσιμες. Με ανησυχεί επίσης το γεγονός ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ε, ε, εντάσσεται σε αυτή την έκθεση και θα πρέπει να το εξετάσουμε, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πρέπει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να παρέχονται αυτές τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλες τις περιοχές και τις αγροτικές. Θα πρέπει, πιστεύω, η Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που είχε η απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδρομείων Και τέλος, καλωσορίζω την άποψη του εισηγητή ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να θεωρηθούν ε, υπηρεσίες κοινής άρα να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά και η δίκαιη τιμολόγηση. Συνολικά πρέπει να πω ότι η έκθεση είναι ισορροπημένη, αλλά θα προτείνουμε και τροπολογίες για να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο στις ε, περιοχές και στα ζητήματα που προανέφερα. Ευχαριστώ. Ε, Vielen Dank. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή ε, ε, συνεργασία, αλλά να ξέρετε ότι εμεί δεν θα την υποστηρίξουμε, θα την καταψηφίσουμε. Και να σας πω και γιατί. Γιατί πιστεύουμε ότι υπησερχόμεθα σε τομεί οι οποίοι, σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, είναι σαφείς ε, ε αρμοδιότητε των κρατών μελών. Και εκεί θα πρέπει να μείνουν. Δεν αποδεχόμαστε λοιπόν αυτή την έκθεση σε ό,τι αφορά τα θέματα που άπτονται του άρθρου 14 των Ευρωπαϊκών Συνθεκών σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία τη Υπηρεσία Κοινή Οφέλεια. Και να διευκρινίσω το εξή, ότι φυσικά θα πρέπει να εναρμονιζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν ποιε είναι οι υπηρεσίε κοινή σε οικονομικού συμφέροντο, πώ θα διοργανωθούν, πώ θα χρηματοδοτηθούν. Φυσικά πάντα τηρουμένων και των ε, κανόνων για τις επιδοτήσεις. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ φοβάμαι ότι η έκθεσή σας θα υπονομεύσει αυτό το σαφές δικαίωμα των κρατών μελών. Και γι' αυτό λοιπόν δεν θα την υπερψηφίσουμε. Γιατί πιστεύουμε κιόλα ότι το γεγονός ότι οι υπηρεσίε κοινή ωφέλεια οικονομικού συμφέροντος διεξάγονται σε επίπεδο ε, κράτους μέλος δεν θα πρέπει να ορίζονται από το εκνητικό επίπεδο. Ισοπαίδωση, ισοπαίδωση είναι αυτή και αυτή προκύπτει σε πάρα πολλέ συζητήσει με του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που το βρίσκουν αυτό παρέμβαση, ανάμειξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο η οικονομική και η χρηματοπιστωτική κρίση, αυτή που μας μαθαίνει σήμερα, είναι και μία κρίση ευθυνών ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι πολίτες να έχουν την εντύπωση ότι δεν χώνει τη μύτη της παντού η Ευρώπη, αλλά ότι γίνεται σεβαστή η επικουρικότητα. Γίνονται σεβαστοί οι νόμοι, οι κανόνες. Αυτό λοιπόν ορίζεται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. είναι θέμα αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης είμαι κατά των λανθασμένων κινήτρων. Να πούμε δηλαδή ότι οι πολίτες οι οποίοι προέρχονται από φτωχά νοικοκυριά, που έχουν άσχημη οικονομική κατάσταση, ότι θα πρέπει να λαμβάνουν δωρεάν κάποιες τέτοιες ε, υπηρεσίες κοινή ωφέλειας. Για παράδειγμα, στο θέμα της ενέργειας, αυτό δίνει ένα λανθασμένο κίνητρο, μια λανθασμένη κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να κάνουν σπατάλες οι πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πιο σωστό θα ήταν να έχουμε για παράδειγμα συσκευέ που θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Όχι να δίνονται τέτοια λανθασμένα κίνητρα. Και επίσης, ποια είναι η Ευρώπη για να ορίσει ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν οι δημόσιε μεταφορές μικρών αποστάσεων. Αν έτσι υποσκάπτουμε την περιφερειακή δημοκρατία, έχουμε μας κάνει εντύπωση αν όλο και πιο μεγάλη είναι η διστακτικότητα των πολιτών έναντι τη Ευρώπης. Όχι, το περιφερειακό επίπεδο είναι θέμα και βάση της δημοκρατίας και της Ευρώπης. Να μην το υποσκάπτουμε και σε ό,τι αφορά το θέμα των αγωγών από πλευρά των ενώσεων. Είμαι αντίθετη. Α, ναι, λοιπόν, θέλετε να αναφέρετε όμως όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλεια, γιατί δεν αναφέρετε και το νερό. Και το νερό είναι τέτοια υπηρεσία. Άρα βλέπετε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ πολιτικά ευαίσθητο θέμα για το οποίο θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Η συνέπεια όμως θα ήταν πραγματικά ότι δεν θα ψηφίσουμε, δεν θα υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση. Ε, Ήρθε και ο κύριος Χατζημαρκάκης, είστε σκιώδης σε αυτό. Ναι, θα ομιλήσω εξ ονόματος του κύριου Σμιτ που είναι ο εισηγητής μας, ο σκιώδης. Θα σας μεταφέρω αυτά τα οποία θα ήθελε να πει. ευχαριστεί τον εισηγητή για την προσπάθειά του, αλλά θα πρέπει να επιλέξει να χρησιμοποιεί τους, τους όρους ευάλωτοι καταναλωτές με μεγαλύτερη ε, προσοχή και επιφυλακτικότητα, γιατί θα απαιτηθεί για αυτές τις κατηγορίες ειδική φροντίδα. Αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά η νομοθεσία δεν είναι ε, ο καλύτερος τρόπος. Η ενέργεια είναι πολύ σημαντικό θέμα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει σε μια πρώτη φάση να εφαρμόσουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις στα πλαίσια της προσπάθειας δημιουργίας μιας πραγματικής αγοράς ενέργειας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ξέρω ότι θέλει ε, και η κυρία Γκέπχαρ το λόγο, αλλά θα ήθελα σαν σκιώδης της ομάδας μου να πω ότι έτσι όπως έχει η έκθεση για διάφορους λόγους δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Εγώ είμαι ευαίσθητος και στα θέματα που έθεσε η κυρία Ρούλε, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Ξεκινώντας θετικά θα έλεγα ότι απαιτείται να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε θέματα τα οποία είναι της αρμοδιότητάς μας. Εδώ η κυρία Γκάλ Πέλτς το έθεσε το θέμα. Η Επιτροπή μας δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σαν παράδειγμα. Το θέμα που μας αφορά είναι το θέμα των καταναλωτών. Υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα σχετικά με τη διαφάνεια και το κόστος της πράσινης ενέργειας και γενικότερα με τα πράσινα προϊόντα και το κόστος τους. Υπάρχουν πακέτα για τους καταναλωτές ε, οικιακής εκμετάλλευσης της πράσινης ενέργειας ε, και αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν, αλλά είναι κυρίως θέματα ε, τα οποία πρέπει να εξετάσουν κυρίως οι συνάδελφοι που ασχολούνται με θέματα αποκλειστικά ενέργειας. Με τις αλλαγές συμπεριφοράς και προτύπων κατανάλωση δεν ξέρω αν ο γνωρίζει τις προηγούμενες εργασίες μας, έχει υπάρξει μια εργασία για τις μεταφορές και για την ενέργεια στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και αυτά τα οποία είχαμε πει τότε παραμένουν σημαντικά και σήμερα. Και γι' αυτό θα είναι καλό να σημειώσετε και κάποια από τα θέματα αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει από λευκό χαρτί. Εδώ ίσως να διαφωνήσουν κάποιοι συνάδελφοι, αλλά λέτε στην εναρκτήρια παράγραφό σας ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με τις ε, υπηρεσίες αυτές κοινή ωφέλεια. Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι υπάρχουν στις, στις ε, ισχύουσες οδηγίες αυτά τα δικαιώματα. Το θέμα είναι να, να εντοπίσουμε καλύτερα, νομίζω, τις υπηρεσίες και η ουσία είναι το τρίτο σημείο σας, ότι ε, επηρεάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή εφόσον γίνονται σεβαστά και εφαρμόζονται τα δικαιώματα του καταναλωτή. Αυτό έχει σημασία. Νομίζω ότι το ύφο της έκθεσής σας και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν διαφωνώ, είναι ότι επιμένετε σε κάποια τμήματα του στα θέματα των δικαιωμάτων σε κάποιους άλλους τομείς όμως ε, απομακρύνεστε λίγο από αυτό και θα πρέπει να επανέλθετε. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να εξετάσετε τη δική μου έκθεση για τις τηλεπικοινωνίες. Οργανώσαμε και χθε μια ακρόαση για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις τηλεπικοινωνίες. Στις τηλεπικοινωνίες συμφωνήσαμε να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο δικαιωμάτων των καταναλωτών λόγω της φύσεως ε, της αγοράς των τηλεπικοινωνιών η οποία ε, δεν θα πρέπει να είναι πολύ, πολύ διασπασμένη. Και θα πρέπει πραγματικά ο καταναλωτής να είναι σε θέση να κάνει τη σωστή επιλογή ανάμεσα σε συγκρίσιμες προσφορές από πλευράς των επιχειρήσεων. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη μορφή της έκθεσης αυτής ήδη διαθέσιμη και νομίζω ότι παράλληλα με τις τηλεπικοινωνίες ε, μπορούμε να διασταυρώσουμε τις προσπάθειές σας με τις δικές μας. Τώρα για τις ταχυδρομικές υπηρεσίε. Η έκθεση του κυρίου Άριας και η ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΚΤ για την παράδοση πακέτων κατοίκων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε έτσι και αλλιώς θέσει τα θέματα της διαφάνειας εδώ, σαν παράδειγμα την ανιχνευσιμότητα του δέματος ε, την πορεία, στην πορεία παράδοσης. Νομίζω ότι απαιτείται μια κάποια εδώ συμβατότητα και θα πρέπει ε, να μην κάνουμε αμφισβητούμενες πολιτικές δηλώσεις. Όπως λέτε σαν παράδειγμα ότι η φιλελευθεροποίηση των ταχυδρομικών αγορών δεν έχουν ωφελήσει τους καταναλωτές. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν εκθέσεις οι οποίες υποστηρίζουν τον ισχυρισμό σας. Αυτή είναι η προσωπική σας άποψη και δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνετε σε μια έκθεση η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα των καταναλωτών. Παρακαλώ να το επανεξετάσετε αυτό. Και στον τομέα των μεταφορών τώρα, η κυρία Ρούλε αναφέρθηκε επίσης και σε άλλους τομείς όπως στους υδάτινους πόρους, τη διαχείριση των υδάτων, και εδώ θα πρέπει να βρούμε περισσότερα στοιχεία για την... Υπάρχουν και τμήματα των μεταφορών, τα οποία δεν αποτελούν τμήμα της παροχής υπηρεσιών κοινή ωφέλεια βέβαια, όπως και τμήματα των μεταφορών και των, της διανομής των ε, ύδατος. Απαιτείται περισσότερη προσπάθεια λοιπόν, θα συνεργαστούμε με χαρά μαζί σας οι συνάδελφοι και θα καταθέσουμε τροπολογίες οι οποίες θα καταστήσουν την έκθεση αυτή αποδεκτή για τη δική μου πολιτική ομάδα, όπως επίσης και για άλλες πολιτικές ομάδες. Κυρία Γκέπχαρτ, έχει το λόγο, δεν ξέρω κάποιος άλλος, κύριος Μάντελ, όχι. Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Ζου, για την καλή συνεργασία. Θα ήθελα να διορθώσω κάποια πράγματα, ωστόσο, για το τι προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Το εξέτασα το κείμενο. Το θέμα δεν είναι να υπησέλθουμε με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο και να ξεπεράσουμε τις ευρωπαϊκές ε, αρμοδιότητες. Θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς οι υπηρεσίε κοινή ωφέλεια ε, προσπαθούν να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Αυτό είναι σωστό ως αρχή και θα ήταν λανθασμένο να απορρίψουμε εξ αρχής μια τέτοια έκθεση. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει αυτή η προστασία. Είδαμε στο παρελθόν ότι σε θέματα ενεργειακής, για παράδειγμα, παροχή σε κάποιες ε, πόλεις στην Τσεχία, στην Πολωνία, ιδιαίτερα το χειμώνα, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό των πολιτών ε, αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν αρκεί να λέμε ότι α, εντάξει, δεν πειράζει, υπάρχουν σε κάποιο επίπεδο κάποιοι κανόνε. Όχι. Ή για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε, κοιτάξτε, λόγω τη απελευθέρωση υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά με του πολίτε. Και προσφάτω έγινε μια πάρα πολύ θελώδη συζήτηση στην Έργη, επειδή σε, μια, σε ένα Δήμο δεν απεστάλησαν τα έγγραφα για συμμετοχή στις εκλογές. Χρησιμοποιήθηκε ένας άλλος πιο φθηνός ε, πάροχος και έτσι, για παράδειγμα, άτομα τα οποία ήταν σε διακοπές δεν έλαβαν τελικά τα έγγραφα αυτά και δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ναι, ναι, κυρία Ρούλη, κοιτάξτε, είναι θέματα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε απλά να πούμε ότι α, να τη σκίσουμε την έκθεση. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε προς τα ποια κατεύθυνση θέλουμε να οδεύσουμε. Τι απαντήσεις θέλουμε να δώσουμε για να διασφαλίσουμε την βασική α, παροχή τέτοιων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Έχει κάποιες καλές προσεγγίσεις η έκθεση. Εγώ, κοιτάξτε, δεν είμαι απαραίτητα υπέρ της ε, ε συλλογικής αυτής ε, αγωγής από πλευράς ε, των ενώσεων γιος, το λέω ξεκάθαρα. Θα το συζητήσουμε όμως και θα κάνω κάποια τροπολογία. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε η προστασία να διασφαλίζεται πραγματικά να διασφαλίζεται. Και πώς μπορούμε να το πατήχουμε αυτό. Δεν είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες ε, γενικού και οικονομικού ε, ενδιαφέροντος και γενής ωφελίας. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δυστυχώς πάρα πολλές υπηρεσίες ελευθερώνονται σε ό,τι αφορά την παροχή τους δηλαδή. Και πολύ απλά και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να φροντίσουμε ότι προστατεύονται τα δικαιώματα του καταναλωτή. κυρία Λάγκια θέλει να παρέμβει. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να... Πρόεδρε, εν συντομία μόνο θα ήθελα να διαφωνήσω με την κυρία Γκέπχαρτ. Φυσικά η απελευθέρωση στον τομέα της, των υπηρεσιών μπορεί να μας βρίσκει αντίθετους, αλλά θα περιοριστούμε σε αυτά που είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Να μην επισέλθουμε στην εθνική αρμοδιότητα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην παρούσα φάση. Προσπαθεί επίπεδος επιστητού σε όλα τα επίπεδα να νομοθετήσει η Ευρώπη και αυτό αυξάνει την αγανάκτηση των πολιτών έναντι της Ένωσης. Και βλέπουμε και στην ομιλία του κυρίου Μπαρόσο στην προηγούμενη Ολομέλεια ότι θα πρέπει να φροντίσουμε μόνο για αυτά τα οποία πρέπει να επιληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αφήσουμε τα εθνικά θέματα σε εθνική αρμοδιότητα. Ε, αυτά τα θέματα είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό ξεκάθαρα και ρητά αναφέρεται στη συνθήκη της Λισαβόνος. Σε αυτά λοιπόν να επικεντρωθούμε. Η ε, κυρία Γκέπχαρτ, μα δεν είπα τίποτα διαφορετικό. Well, Mr. also was hoping for a lively debate, so we certainly had one so far ζητήσατε να κάνουμε μια συζήτηση και από ό,τι βλέπω ήδη ξεκίνησε μια ζωντανή συζήτηση. Φαντάζομαι ότι οι συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών θα είναι εξίσου δυναμικές. Θα έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας. Ας ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Ε, μετά θα ακούσουμε την κυρία Ποτσμάσκη. Επομένως δίνω το λόγο στην κυρία Μπλουμ την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρία Βάιντενχολτσε. Πρώτα απ' όλα να, σας, να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Επίση, ευχαριστούμε και τους βουλατές αυτές που τοποθετήθηκαν σήμερα το πρωί. Όπως γνωρίζετε, από τον Ιούλιο υπάρχει ένας επίτροπος, ο κ. Νίμιτσα, ο οποίος είναι αρμόδιο για τα ζητήματα προστασίας του καταναλωτή. Και το γεγονό ότι υπάρχει ένας επίτροπος αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά ε, καταδεικνύει την ε, σημασία που τους αποδίδουμε, ιδίως σε μια περίοδο κρίσης. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, ο Επίτροπος Νίμιτσα έχει υπογραμμίσει τη σημασία οι καταναλωτέ να έχουν στη διάθεσή τους πιο οικονομικές υπηρεσίες σε τομείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές που αναφέρονται και στη γνωμοδότηση Αναγνωρίζουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η γνωμοδότηση καλύπτει πολλές, πολλούς, πολλά θέματα. Ορισμένα είναι τομεακά, ορισμένα είναι ε, οριζόντια, κάποια, και αναφέρθηκε αυτό, δεν ρυθμίζονται ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την ε, γνωμοδότηση και μπορώ να σας ενημερώσω ήδη ότι για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας, του οποίου η σημασία έχει τονιστεί, Στον τομέα λοιπόν της ενέργειας θα σας παραπέμψω στο έργο που έγινε στο πλαίσιο του Φόρουμ ε, των Πολιτών για την Ενέργεια και στο τρίτο πακέτο για την ενέργεια. Στις 16 Δεκεμβρίου προετοιμάζουμε τις εκθέσεις ε, της συζήτησης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, δηλαδή τη συζήτηση που διεξήγε η Επιτροπή με τις εποπτικές αρχές, τον κλάδο, τη βιομηχανία, και τις οργανώσεις καταναλωτών. Και οι εκθέσεις αυτές συνδέονται με δύο θέματα που αναφέρονται στη γνωμοδότησή σας. Πρώτα απ' όλα την ηλεκτρονική τομολόγηση και την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Και επίσης το ζήτημα της διαφάνειας των τιμών, της τιμολόγησης και της συγκρισιμότητας της τιμολόγησης. Θέματα τα οποία έχετε φίξει στη γνωμοδότησή σας. Επίσης η δεύτερη έκθεση αναφέρεται στους, καταναλωτές, στους ιδιαίτερα ευάλωτους καταναλωτές. Και αυτά, αυτές οι δύο εκθέσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη συζήτησή μας με την Επιτροπή. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά, γιατί υπάρχει ήδη μια νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής, η ΣΑΝΚΟ και άλλες, συνεργάζονται και εργάζονται σκληρά έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι η φυστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία εφαρμόζεται και συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη. Στόχος μας λοιπόν με αυτές τις εκθέσεις είναι να καταγράψουμε τις βέλτικες πρακτικές έτσι ώστε ε, εάν υπάρχει μια ε, πρακτική η οποία λειτουργεί καλά σε κάποιο κράτος μέλος αυτή να χρησιμοποιηθεί και από τα υπόλοιπα για να επιταχυνθεί και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά και έχουμε τα στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό, ότι η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος, σε κράτος μέλος. Αλλά πάντως η ενέργεια είναι ένας τομέας στον οποίο οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιημένοι από τη σημερινή κατάσταση. Έρχομαι τώρα στις τηλεπικοινωνίες προετοιμάζεται μια πρόταση της Επιτροπής, μια πρόταση πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες που ευελπιστώ ότι θα αντιμετωπίσει και κάποια από τα θέματα που φύγετε στην έκθεσή σας. Αλλά υπάρχουν και άλλες θεματικές που πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Έχουμε ξεκινήσει μια μελέτη ε, στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ για τους ευάλωτους καταναλωτές και εδώ εστιάζουμε περισσότερο σε νέο, νέα είδη ε, ευάλωτων καταναλωτών, νέες μορφές ευάλωτων καταναλωτών. Με όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα σας ε, βοηθήσουμε στη συζήτησή σας και δίνω το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Μάρκτ. Ο Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να ζητήσω να προσέχουμε, να, να, να, να σεβαστούμε λίγο τους ε, προσκεκλημένους μας και ε, εάν είναι απαραίτητο να κάνετε κάποια συζήτηση μπορεί να γίνει εκτός της αίθουσας αυτή για να είμαστε ήσυχοι εδώ. Κύριε Σποτσμάρσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Εγώ κυρίως θα αναφερθώ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αναφέρεται στην έκθεσή σας ότι πρέπει να διασφαλίζεται η γενική ταχυδρομική υπηρεσία σε ολόκληρη την επικράτεια μιας χώρας με λογικές τιμές και λογική ποιότητα με βάση μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δηλαδή όλες εκείνε οι οποίε καταγράφονται στην οδηγία για τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε, ε, είναι πλήρως διασφαλισμένες και στα 28 κράτη-μέλη. Ξεκινήσαμε με την πράσινη βίβλο και έχουμε εξετάσει το ζήτημα των ταχυδρομικών υπηρεσιών με συνεκτικό τρόπο. Η οδηγία έχει τις αιτιολογικές 19 19-2021, ε, στις οποίες αναφέρεται η σημασία των παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές. Πρέπει βεβαίως να διασφαλίσουμε την εφαρμογή στην πράξη αυτής της ε, νομοθεσίας. Το άρθρο 19 της οδηγίας προβλέπεται μια διαδικασία ε, προσφυγών σε περίπτωση που δεν υπάρχει ε, σωστή εφαρμογή των ταχυδρομικών υπηρεσιών, σωστή παροχή αυτών των υπηρεσιών. Και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, η οδηγία αναφέρει ρητά ότι οι εποπτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν σε περίπτωση παραβίασης των συνθήκων εργασίας. Και αυτό είναι ουσιώδης ε, απέτηση. Η οδηγία είναι σαφής ως προς αυτό και θα έλεγα ότι είναι καινοτόμο στοιχείο της. Η οδηγία μάλιστα είχε εγκριθεί με ευρύτατη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάνω από 500 μέλη την είχαν υπερψηφίσει. Στο ζήτημα τώρα τη απελευθέρωση των, ε, ε, ε, υπηρεσιών αυτών δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι η απελευθέρωση οδήγησε σε άσχημα αποτελέσματα. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι η απελευθέρωση κατάφερε τα πάντα όσο θα θέλαμε και βεβαίω υπάρχουν και διεστάμενε απόψει. Τα επόμενα χρόνια η Επιτροπή δημιουργεί μια διαδικασία, μια έκθεση, η οποία θα αξιολογεί με αντικειμενικό τρόπο τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης. Δεν θα είναι η κατάσταση δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Είναι κάπως ενδιάμεσα τα πράγματα. Κάποια στοιχεία είναι θετικά, κάποια αρνητικά. Τώρα, α μην ξεχνούμε επίση ότι ο Επίτροπος Μισελ Μπαχνιά είχε δημιουργήσει το Φόρουμ Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, στα οποία ε, συμμετέχουν εκπρόσωποι των Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, οι ταχυδρομικοί πάροχοι, υπηρεσιών, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η ΕΟΚΕ επίσης αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος και θα το εξετάσουμε και στην έκθεση εφαρμογής που προετοιμάζουμε. Είναι μια υπηρεσία η οποία αφορά πάρα πολλούς πολίτες. Αναφέρεται στην παράδοση της αλληλογραφίας μας καθημερινά, παντού στην Ευρώπη. Οι ταχυδρομικέ υπηρεσίε αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας. που είναι προ το συμφέρον όλων μας να είναι επαρκής. Και θα εξετάσουμε, όπω είπα, το ζήτημα στο, στην έκθεση που προετοιμάζουμε. Τώρα η Επιτροπή επίσης πριν το τέλος του 2013 προετοιμάζει μια έκθεση για την ε, ολοκληρωμένη δρομολόγηση. Και επίσης το γεγονός ε, ε, του σεβασμού των συνθηκών εργασία Και αυτό το θέμα το θεωρούμε σημαντικό. Εδώ δεν αναφερόμαστε κυρίως στους ε, παρόχους γενικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Εκείνοι σέβονται αυτά τα δικαιώματα και τις εργασιακές συνθήκες. Το ζήτημα είναι με άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Γνωρίζουμε τέτοια περιστατικά από τον τύπο. Σε, σε, σε εταιρείες ε, υπεργολάβους, ορισμένες εταιρείες λοιπόν παραβιάζουν αυτά τα εργασικά δικαιώματα. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα ότι στη συμφωνία για την κυβέρνηση της συνεργασίας στη Γερμανία καταγράφεται ως ε, στοιχείο της συμφωνίας ότι οι τιμές ε, των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Γερμανία θα παραμείνουν σταθερές. Βλέπετε λοιπόν πόση σημασία αποδίδουν σε αυτά τα θέματα και τα κρατημέλη. Την επόμενη χρονιά λοιπόν ε, θα έχετε στη διάθεσή σας την ε, έκθεση και θα μπορέσετε να την αξιοποιήσετε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τόμπρον και την κυρία Πουτίνσκι που βρέθηκαν εδώ και μας βοηθήσαν να εντοπίσουμε κάποια από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Να δώσω στον κύριο Βίνχολτς την ευκαιρία να απαντήσει εν συντομία όμως, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες και να μας παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει καταστεί σαφές ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, έχει και πάρα πολύ θόρυβο άλλωστε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σημαντική συζήτηση που έγινε, τα σημαντικά, τις σημαντικές παρατηρήσεις και προσβλέπω σε μια πιο εντατική συζήτηση. Νομίζω ότι αποδέχτηκε σήμερα ότι το θέμα είναι αρκετά αμφιλεγόμενο και χρήζει επισταμένη συζήτηση. Αυτό πρέπει να γίνεται στο Κοινοβούλιο, το ελπίζω δηλαδή. Από τη ζωντανή συζήτηση ελπίζω να προκύψει και μια καλή έκθεση. Γι' αυτό ζητώ από όλους τους συναδέλφους να μην τοποθετούνται τόσο αρνητικά και απόλυτα εξ αρχής κυρία Ρούλε να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Ένα μόνο επιχείρημα θα ήθελα να προτάξω. Στη συζήτηση πιο πολύ, πιο λίγη Ευρώπη, όταν ξέρει κανείς ότι κάποιες ε, αρνητικές καταστάσεις προέκυψαν από ευρωπαϊκή παρέμβαση, νομίζω ότι ενδεχομένω να χρειάζεται και ευρωπαϊκή παρέμβαση για να τα περιορίσει κανεί ε, αυτά τα αρνητικά στοιχεία τα οποία προκλήθηκα από την Ευρώπη. Αυτά θα τα συζητήσουμε στα πλαίσια τη συνεδρίαση των σκιωδών. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Well, I agree with you. Θα συμφωνήσω μαζί σα. Πράγματι ήταν καλή συζήτηση μέχρι τώρα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα και θα επανέλθουμε στα επιμέρους θέματα που τέθηκαν σήμερα το πρωί. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η 10η Δεκεμβρίου. Θα εξεταστούν στη συνεδριάσή μας στις 22 και 23 Ιανουαρίου και θα ψηφίσουμε στις 11 Φεβρουαρίου για να φτάσουμε στην Ολομέλεια πριν από τις εκλογές. Περιμένω λοιπόν το πως θα καταλήξει η τελευταία από τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες φορές στην πολιτική συζήτηση ευρύτερα. Θα συνεχίσουμε τώρα με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Ευχαριστώ κυρίως τους αντικαταστάτες, αναπληρωτές. Θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε να μην βαρεθείτε. Ελπίζω να έχετε όλη την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας. Απαιτείται αυτό. Σήμερα θα ψηφίσω και εγώ εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Η πρώτη έκθεση είναι μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών για τις ηλεκτρονικές κλήσεις, το e-call, Ξέρετε ότι στο τέλος της συνεδρίασης, μετά την ψηφοφορία, θα έχουμε εμείς ε, ε, μια παρουσίαση ενδιαφέρουσα της εφαρμογής του συγκεκριμένου συστήματος e-call στα πλαίσια του συστήματος ε, ηλεκτρονικής πλοήγησης, δορυφορικής πλοήγησης, αυτοκίνητα δηλαδή. Η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα αλλά απαιτείται να στείλουμε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Μεταφορών έτσι ώστε να συμβαδίζουμε χρονικά μαζί της. Δεν ξέρω αν έκανα κάποιο λάθος, η κυρία Σενάλοβα θα με διορθώσει. Λοιπόν, ψηφίζουμε στο άρθρο 1, στον τίτλο της έκθεσης, δηλαδή ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 11 έχει αποσυρθεί. Η 12. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία του κυρίου Βάιντερ Χόλτζερ. Γίνεται δεκτή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Αμέσως μετά πηγαίνουμε στην 4, στην τροπολογία 4. Α, όχι, συγγνώμη, ξέχασα την τροπολογία 3, λέει ο πρόεδρος. Ένα νέο ένα 1α μικρό. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε μετά στην τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Δεκτή και αυτή. Τώρα ξεκινάει η ψηφοφορία. Θα μετρήσουμε πρώτα τους ψηφίζοντες. Στο σύνολο του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία. 32 ψηφίζουν. 32 κανονικά ψηφίζουν. 34. Λοιπόν, κάποιος που δεν ψήφισε. 34 κάρτες λοιπόν. Πέρα της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 5 κατά και 0 αποχές. Ευχαριστώ την κυρία Σενάλοβα. Περνάμε τώρα στην έκθεση του Σέρτζο Κοφεράτη. Μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αν δεν κάνω λάθος, για τη σωστή ενημέρωση σχετικά ε, με τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις στο μη χρηματοοικονομικό τομέα. Θέλετε κάτι να πείτε εισαγωγικά κύριε Κοφεράτη, όχι. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 36. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψήφος εδώ για την 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ να ψηφίζετε λίγο πιο γρήγορα. Υπάρχει μία κάρτα ακόμα που δεν ψήφισε, εν πάση περιπτώσει, η μία κάρτα που δεν ψηφίζει να ψηφίσει γιατί μπορεί να είναι αποφασιστική η ψήφος αυτή. Λοιπόν, γίνεται δεκτή. Η 37. Εδώ υπάρχει μία προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή και αυτή. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Α, συγγνώμη. Εδώ υπάρχει και χωρισμένη ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτό. Συμβιβαστική 2. Στη συμβιβαστική τροπολογία 1 το δεύτερο τμήμα. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας 16 υπέρ, 17 κατά απορρίπτεται. Οπότε καταπίπτουν αρκετές άλλες τροπολογίες. Και πηγαίνουμε στη σελίδα 4, στην τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 56 καταπίπτει. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή και αυτή. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 14 το εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 14. Τέλος της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή. Η τροπολογία 60 τώρα, ψηφίζουμε την 60. Τέλος. Απορρίπτεται. 61 με προφορική τροπολογία του εισηγητή ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 1α μικρό. Είχε γίνει δεκτή βέβαια μέσω της τροπολογίας 1 αυτή. Πηγαίνουμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις, στην τροπολογία 24. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 4, υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 5, υπέρ, κατά, δεκτή. 29, υπέρ, κατά, δεκτή. 30, υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, δεκτή. 33 υπέρ, κατά, δεκτή. 34 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, δεκτή. Οπότε αρχίζει η ψηφοφορία τώρα για το σύνολο της προτάσεως ψηφίσματος όπως τροπολογήθηκε. Okay. So 33 cards in. Right, the vote's closed. Πέρα της ψηφοφορίας, 29 υπέρ, 3 κατά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κοφεράτη. Ε, Καλώς τώρα θα περάσουμε στην συνολική έκθεση του κυρίου Χατζημαρκάκη Θα θέλατε να κάνετε μια εισαγωγική παρατήρηση κύριε Χατζή όχι. Ε, let's start the vote. Ε, ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Στην τροπολογία 1 του τι υπέρ της 1 κατά δεκτή. Η 55 καταπίπτει. Συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 20 υπέρ. Η 20 5 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 30 υπέρ κατά δεκτή. Η 6 συμβιβαστική υπέρ κατά δεκτή. Η 13 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά δεκτή. Η 14 ε, νομίζω ότι είναι τεχνική αλλαγή. Υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, δεκτή. 16 του εισηγητή υπέρ, κατά, δεκτή. Η 7 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 10, υπέρ, κατά, δεκτή. Η 20 τεχνική τροπολογία. Περνάμε στην 23. Εδώ υπάρχει και χωρισμένη ψηφοφορία ζητήθηκε από τους σοσιαλιστές. Το πρώτο τμήμα της 23 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη. 16 υπέρ 16 κατά. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν έχει καταπέσει επειδή απερίφθη το πρώτο. Τώρα περνάμε στην 124 του κυρίου Τσαρσκόφσκη. Α, έχει καταπέσει και αυτή. Περνάμε στη συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Απασχόληση 24. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες απερίφθη. Απασχόληση 25. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απερίφθη. 26 και 27 132 με προφορική υπέρ. Κατά. Νομίζω θα πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα στις ψηφοφορίες είχε πράγματι απεριφθεί. 16 υπέρ, 16 κατά. Πάντως καλά κάναμε και ελέγξαμε, λέει ο Πρόεδρος. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 16. Κατά. Δεκτή. Η 137 καλύπτεται. Η 25 είναι τεχνικής φύσεως αλλά πρέπει να την ψηφίσουμε. 25 υπέρ κατά δεκτή. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά δεκτή. Περνάμε τώρα στην 26 του εισηγητή υπέρ, κατά δεκτή. Απασχόληση 30 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας επιπλέον φαίνεται να ψηφίζει πέρα ψηφοφορίας. Απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. Περνάμε λοιπόν τώρα. Έχει καταπέσει 143, 146 αποσυρθεί. Περνάμε στην 147 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική 21 έχει ήδη καλυφθεί από την προηγούμενη συμβιβαστική. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα τις 158. Πιατικά είναι. Άρχεται η ψηφοφορία για την 158. Πέραστη της ψηφοφορίας απερίφθη. Απασχόληση 31. Άρχεται η ψηφοφορία για την 31. Τέλος. Δεκτή με μία ψήφο διαφορά. Συμβιβαστική 22 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 164 υπέρ. Ηλεκτρονική ψήφος παρακαλώ για την 164 ελέγχουμε. 19 υπέρ, 14 κατά τελικά δεκτή. Η 162 απεσήφη, 25 υπέρ, κατά δεκτή. Απασχόληση 33 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 34 δεν τίθεται σε ψηφοφορία. so it's better to have the vote here and to indicate that the block is consistent of amendments 30, 34, 35, 37. Right. We're voting on all okay. Okay. So uh, we've just come now to a. Φτάσαμε τώρα σε μια ομαδική ψήφο, η οποία καλύπτει και τον τίτλο. Τίθεται σε ψηφοφορία λοιπόν τροπολογίες 34, 35 και 37. Εντάξει. 34, 35 και 37. Λοιπόν. Προηγείται των υπολείπων ομαδικών. Έτσι κι αλλιώς παραμένει συμβιβαστική τροπολογία, απλά έχει αλλάξει η σειρά για να γίνει πιο λογικό αν γυρίσετε σελίδα θα δείτε 34 και 37, 35 και 37 δεν είναι σε συμβιβαστική. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτές. Συμβιβαστική 23 υπέρ, κατά, δεκτή. Αν γυρίσετε τη σελίδα θα δείτε ότι ψηφίσαμε το 34 και 35. Περνάω λοιπόν στην 24. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα την 183 υπέρ τα δεκτή. Η 37 ψηφίστηκε, περνάμε στη συμβιβαστική 26 υπέρ κατά δεκτή. Επανέρχομαι στην 39 του εισηγητή υπέρ κατά δεκτή. Πολιτισμός 13 υπέρ έχει καταπέσει. Απασχόληση 35. Άρχεται η ψηφοφορία για την απασχόληση 35. Λοιπόν, τώρα έχουμε 34 που ψηφίζουν απερίφθη. Η 35. 187 έχει καταπέσει. Οπότε πηγαίνουμε στην 29 πλέον, συμβιβαστική 29. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τώρα πηγαίνουμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Η 56. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Κατά. Δεκτή. Τώρα η 2 και η απασχόληση 2 έχει γίνει αυτόματα δεκτή με την προηγούμενη τροπολογία. Η 58 έχει καταπέσει, η 57 έχει καταπέσει, ο πολιτισμός 1 έχει καταπέσει, 59 έχει καταπέσει, φτάνουμε στην 60. Η 60 λοιπόν, Μωράες, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Προφορική τροπολογία, ποιοι είναι υπέρ κατά, δεκτή. 61 υπέρ, κατά, δεκτή. 62 καταπίπτει. Συμβιβαστική 1, ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτή. Πολιτισμός 2. Πολιτισμός 2, ποιοι είναι υπέρ, Πέρα της ψηφοφορίας. Μία ψήφος διαφορά δεκτή. Η 64 καταπίπτει. Απασχόληση 5 καταπίπτει. Η 6 αυτόματα δεκτή. Η 65 απαράδεκτη. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. 67 και απασχόληση 7 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 68. Πολιτισμός 3. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πολιτισμός 4. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η τροπολογία 70 και απασχόληση 8. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε. 70 και 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Υπάρχουν πολλές κάρτες που δεν ψήφισαν. Πέρα της ψηφοφορίας δεκτή. 19 υπέρ 15 κατά. Ψηφίζουμε τώρα την 69 που είναι συμβατή. 69. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Πολιτισμός 5. Αρχίζει η ψηφοφορία για τον πολιτισμό 5. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 18 υπέρ 15 κατά. Απασχόληση 9. Έχει ήδη καλυφθεί. Δεν την ψηφίζουμε. Πηγαίνουμε τώρα στον πολιτισμό 7. Όχι, για μια στιγμή λέει ο Πρόεδρος. Ελέγχομαι το τι θα κάνουμε με την 72. Uh, λοιπόν, η 72 είναι συμβατή και δεν καλύπτεται, οπότε την ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, δεκτή. 7. Ποιοι είναι υπέρ κατά, δεκτή. Η τέσσερα έχει ήδη καλυφθεί, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε τον πολιτισμό 8. Άρχεται η ψηφοφορία για πολιτισμό 8. Έχουμε φτάσει στην 35. Μία ψήφος διαφορά 18 υπέρ 17 κατά. Η 73 καταπίπτει. 74 του κυρίου Βάιντεν Χολτσεφ. Ποιοι είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. 35 η ψήφοι. Εγκρίνεται. Τη απασχόληση 11 υπέρ. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναξη ψηφορίας. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Να ψηφίσουμε την 75. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Μέσα ψηφία. 12 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ένα ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 13 της Επιτροπής Απασχόλησης. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Η 77 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78. Εγκρίθηκε. Η 14 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναξη ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Προχωράμε στην 15 της Επιτροπής Απασχόλησης σε δύο τμήματα που έχει ζητηθεί από τους Σελδημοκρατές. Πρώτο τμήμα λοιπόν, ένα ψηφορίας. Για την 15 της Επιτροπής Απασχόλησης, πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα λοιπόν στην 15 της Επιτροπής Απασχόλησης. Καταπίπτει λοιπόν το δεύτερο τμήμα. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, γιατί έχει καλυφθεί από προηγούμενη ψηφοφορία. Και η 80 καταπίπτει, επειδή πέρασε η συμβαστική 17, αλλά μπορούμε να την ψηφίσουμε προσθήκη. Η 80 ως προσθήκη λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 6. Καταπίπτει η 81 ή 82 λοιπόν. Η 82. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, 17 κατά. Η 83 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Η 84, η 84, λυπάμαι. Η 84, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 92. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 17 της Επιτροπής Απασχόλησης επίσης. Η 8 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 93 κατά πίπτη. Α, μάλιστα. Ε, η συμβαστική 23. Η 95 συμβατή. Ως προσθήκη. Η 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στα παρατήματα. με τη συμβαστική 5 γίνεται αποδεκτό όλο το τμήμα για τα παρατήματα. Πολύ ωραία. Και περνάμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα, Block B, σελίδα 32 στον κατάλογο ψηφοφορίας, συμβιβαστική 27, σε τέσσερα τμήματα. Εντάξει, το βρήκατε όλοι. Η συμβιβαστική 27 σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. The vote's closed. Πέρας. Πάρα πολύ γρήγορη. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Γρήγορα, γρήγορα, παρακαλώ. Εγκρίνεται με τρει ψήφου διαφορά. Τέταρτο τμήμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν καταπληκτούν. Όλο το παράτημα. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία τώρα. Έναρξη ψηφοφορίας για το σύνολο της έκθεσης. Yeah, okay. Well, I'll give the report to the rapporteur first. Uh, are there two more people who want to vote on this or not? Άλλοι δύο θέλουν να ψηφίσουν. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 30 ψήφοι υπέρ, κατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζημαρκάκη. Νομίζω Λίγη ησυχία παρακαλώ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή. Πώς σκοπεύετε να ανταποκριθείτε, να απαντήσετε και ποιες είναι οι προοπτικές μας να συνάψουμε συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, ποια στρατηγική θα ακολουθήσει με τους κοιόδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η νομοθεσία, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική, τουλάχιστον για 10% του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά προσβασιμότητα ιστοσελίδων για κοινές, ε, κοινοφελείς υπηρεσίες. Έχουμε λοιπόν ένα στόχο, αν θέλουμε, ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Το Συμβούλιο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει το θέμα των συζητήσει στην ομάδα εργασία το Δεκέμβριο η Λιθουανική Προεδρία. Μα είπαν ότι θα το κάνουν. Η Ελληνική Προεδρία, οι Έλληνε, σε έναν τριμερή διάλογο τον Γενάρη θα προσπαθήσουν να πετύχουν συμφωνία μαζί μα. Είναι εφικτό αυτό. Συζητήσαμε το θέμα αυτό ήδη με την Προεδρία. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή, ακλόνητη θέση του Κοινοβουλίου που θα επιτρέψει στην Ελλάδα στου Έλληνε, να το εξετάσουν αυτό, να κάνουν ενδεχόμενε διαπραγματεύσει, να κάνουν ενδεχόμενου συμβιβασμούς, γιατί στο ιστορικό του Συμβουλίου το Φεβρουάριο θα γίνει η ψηφοφορία είτε στην, πρώτη, στην δεύτερη ολομέλεια του Στρασβούργου θα γίνει η ψηφοφορία και μετά θα ολοκληρωθεί λοιπόν με τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ που δώσαμε τέτοιο ηχηρό μήνυμα με την ισχυρή πλειοψηφία. Ναι, Ωραία. Έγινε λοιπόν κάποια σημαντική πρόοδο, λέει ο πρόεδρο, Θα πρέπει να δοθεί επισήμω η εντολή τον Δεκέμβριο, αλλά προφανώ εσεί και οι σκιώδες συζητητέ θα μπορέσετε να κάνετε ανεπίσημε συζητήσει ήδη και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Αν ακολουθήσετε, αν πετύχετε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προφανώ αυτό θα σημαίνει Απρίλιο μετά. Να είμαστε έτοιμοι. Θα το αποφασίσει λοιπόν η γραμματεία αυτό γιατί υποπτεύομαι ότι θα προσπαθήσουν γρήγορα γρήγορα να προσθέσουν διάφορα στοιχεία και οι άλλες επιτροπές. Θα είναι και πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία στην Ολομέλεια. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν με τη γραμματεία, τη στρατηγική. Το Μάρτιο θα είμαστε καθυστερημένοι, καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε και την cooling off phase. Το Φεβρουάριο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτά επειδή έχουμε δύο ολομέλειες, ξέρετε, νομίζω ότι ο Πρόεδρος για τη στρατηγική σας θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει, να την υποστηρίξουμε. Ελπίζουμε να πετύχετε τη συμφωνία με το Συμβούλιο, προκειμένου να έχετε το τελευταίο κείμενο, το τελικό κείμενο, και αυτό να υποβληθεί στην Ολομέλεια. Αυτή νομίζω ότι είναι η στρατηγική. Αν είναι ένα νομοθετικό κείμενο που θα συμφωνηθεί με το Συμβούλιο και μου αποσταλεί μία επιστολή και μου πούν ότι κοιτάξτε, συμφωνεί το Κοινοβούλιο, αυτό θα σήμαινε δύο μήνες. Άρα στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπολογίσετε τον Απρίλιο. Προφανώς το κείμενο είναι αρκετά περίπλοκο. Αυτό θα είναι μία απόφαση που θα πρέπει να τη λάβετε μετά την πρώτη, τον πρώτο γύρο συζητήσεων με το Συμβούλιο για να δείτε ποιες θα είναι και οι προοπτικές σας. Είναι σαφέ αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εντελεχώ να το συζητήσουν αυτό οι συντονιστές καθότι πρόκειται για δικαίωμα των πολιτικών ομάδων. Άρα μπορείτε να κάνετε εσεί την πρόθεσή σα, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί και αναλόγω. Και θα πρέπει να σας καλέσουμε αν σημειωθεί αυτή η πρόοδος στους συντονιστές με πλήρη υποστήριξη όλων των σκιωδών προκειμένου να υποβάλλετε την πρόστασή σα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα. Uh, Ο κύριος Σφάπ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές σήμερα το πρωί, αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσουν και τους κοιόδης εισηγητές σε ό,τι αφορά την τελική ψηφοφορία για την έκθεση Χατζημαρκάκη. Το είπατε και χθε ο κύριος Συνάδελφο Κατσόφσκι από τον, Υπουργείο Ψηφιακής Ατζέντα της Πολωνίας ε, κλήθηκε και χαιρόμαστε ω ΕΛΚ που συμμετείχε. Του ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία και ελπίζουμε να συνεχίσει τις εργασίες τους στη νέα του ιδιότητα σε ό,τι αφορά το Πολωνικό Υπουργείο που θα αναλάβει. Well, I'm really delighted that uh, Rafael Draskowski has managed to join us on his way to important duty. Χαίρομαι λοιπόν που μπόρεσε να έρθει εδώ και θα μας λείψει από την Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά, ε, παρ όλα αυτά πρέπει να σας συγχαρώ για τον νέο σας ε, πόστο. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την εκθέση για την προσβασιμότητα, <laughs> μπορείτε να γνωρίζετε ότι τουλάχιστον ένα κράτος μέλος θα την υποστηρίξει και θα υποστηρίξει την προσπάθεια να την ολοκληρώσουμε γρήγορα. Πάντως πρέπει να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια της καλής συνεργασίας που είχαμε και ελπίζω να μην χαθούμε. Ε, από την πλευρά μου θα το επιδιώξω πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ξαναμιλήσουμε σύντομα. Έχουμε ακόμα μια ψηφοφορία τεχνικής φύσεως. Για, τον... για τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών. Πρέπει να σας ενημερώσω και για τα πρακτικά ότι ψηφοφορία που είχαμε στο σημείο 19 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υποπίεση έχει αναβληθεί. Γιατί το θέμα συζητείται στο Συμβούλιο και νομίζω ότι εδώ είναι ε, η πρώτη φορά που θα κάνουμε ψηφοφορία. Τώρα στο θέμα 20 ε, για τον τομέα των δομικών έργων. Ήταν πολύ περίπλοκο ο φάκελο που η κυρία Στάιλερ πραγματικά τον εξέτασε εντελεχώ. Σα δίνω λόγο για να ε, παρουσιάσετε αυτό που θέλετε. Είναι μία και μοναδική ψηφοφορία για να εγκριθεί. Δεν μπορεί να ε, τροποποιηθεί. Μπορούμε μόνο να το εγκρίνουμε ή να το καταψηφίσουμε. Έχετε λοιπόν το λόγο για να μας παρουσιάσετε και να δούμε αν συμφωνούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία ήταν ενδιαφέρουσα και οι σκιώδεις εισηγητές ε, είχαμε με, με αυτούς μια πολύ καλή συνεργασία. Όπως είπατε, μπορούμε απλώς να υπερψηφίσουμε, να καταψηφίσουμε. Η πρότασή μου είναι να την υπερψηφίσουμε. Η διαδικασία ήταν μακρά, αλλά νομίζω ότι τελικά το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο δυνατό για το μέλλον. Ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε και κυρίως, σε σχέση με την τεκμηρίωση ε, των ιστοσελίδων, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να βελτιώσουμε στο μέλλον την νομοθεσία. Κάναμε μια συζήτηση σχετική με το, την Επιτροπή και τους ε, Σκιώδης. Πάντως, ο κανονισμός που έχουμε αυτή τη στιγμή επιτάπητος ε, είναι νομίζω προς τη σωστή κατεύθυνση και ζητώ από τους συναδέλφους να τον υπερψηφίσουν. Ο Πρόεδρος θέλει κάποιος άλλος μήπως το λόγο. Κυρία Ρούλε. πολύ σύντομα να τονίσω ότι περιμένουμε από την Επιτροπή να καταθέτει τέτοιου τύπου τη της πράξης εγκαίρως. Ο τομέας των δομικών έργων το περίμενε ήδη από τον Ιούλιο και Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτή τη συζήτηση και αυτή τη ψηφοφορία, γιατί ε, ο τομέα, ο κλάδο έπρεπε να κάνει τι σχετικέ ε, διατυπώσει. Και θα ψηφίσουμε επιτέλου τώρα για κάτι, αλλά θα ήταν καλύτερο να το είχαμε ψηφίσει πολύ νωρίτερα. Πρόεδρος. Ε, ναι, έχετε δίκιο και πράγματι στο ψήφισμα έχουμε συμπεριλάβει ένα σχόλιο σχετικό για την καθυστέρηση από την πλευρά της Επιτροπής και σωστά αναφέρατε ότι ο τομέας των δομικών έργων ανέμενε με ανυπομονησία αυτόν τον κανονισμό. Συμφωνείτε και εσείς, κυρία Στάιλερ, ε, και είχαμε μια, την, την ίδια συζήτηση για τον εξοπλισμό υποπίεση. Και εκεί θα έπρεπε να κινηθούμε πιο γρήγορα. Το λέω αυτό μπα και μας ακούει κανένα από το, μέσω ίντερνετ από το Συμβούλιο. Με πάση περιπτώσει, προχωρήσουμε με, τις, ε, με τα δομικά έργα. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την κατεξουσιοδότηση πράξη για τις δηλώσεις απόδοση προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που διατίθενται σε ιστοσελίδα. 28 παρόντες ψήφισαν όλοι, όχι 31 είναι ανοιχτή η ψηφοφορία ακόμα. Λήξη ψηφοφορία τώρα. 29 υπέρ, ένας κατά, ε, τέλος πάντων. Με ξεκάθαρη πλειοψηφία εγκρίνεται. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σας για την ε, ψηφοφορία. Ήταν πολύ ε, αποτελεσματικές οι συμβαστικές τροπολογίες. Ο προσκυκλισμένος μας για το σημείο 21 θα έρθει στις 11. Επομένως, κυρία Στεράλαβα, δεν ξέρω αν μπορούμε να συζητήσουμε από τώρα. Πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Είχαμε προβλέψει τόσο χρόνο για την ψηφοφορία, γιατί πιθανόν να έπαιρνε περισσότερο με τις συμβαστικές τροπολογίες. Εν πάση περιπτώσει, διακόπτουμε μέχρι τις 11.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 Uh, so, um, uh, Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά. Περνάμε στο τελευταίο θέμα σήμερα, που είναι μια ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκομένους για το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την ανάπτυξη του συστήματος e-call και τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Είχαμε ήδη μια συζήτηση με την κυρία Σενάλοβα Όσοι είσαστε εδώ ξέρετε ότι ξεκινήσαμε και με μία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας εδώ και 1,5 χρόνο. για να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Πολλά έχουν μεσολαβήσει από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό το 2003 και με χαρά βλέπω ότι φτάνει στην τελική φάση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν σήμερα είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους από τους βασικούς εμπλεκομένους να εκφραστούν και να ασχοληθούμε με κάποια από τα θέματα τα οποία αφορούν και τις τροπολογίες τις οποίες καταθέτουμε στην πρόσταση, κυρίως το θέμα της προστασίας των δεδομένων, τη διαθεσιμότητα του Γαλιλαίου και το τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από τα πιλωτικά προγράμματα που είναι πολύ σημαντικά έτσι ώστε να πισθούν τα εναπομείναντα κράτη-μέλη που διστάζουν. Γνωρίζετε και δεν το κρύβω αυτό ότι υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες δεν είναι απόλυτα ακόμα πεπισμένες για τις ε, ικανότητες που έχουν τα συστήματα αυτά για να διασώζουν ανθρώπινες ζωές σε σχέση με το υψηλό τους κόστος. Αυτό θα θέλαμε λοιπόν να το ε, εξετάσουμε. Κάνουμε προσπάθεια για να πείσουμε με την ε, σκληρά εργαζόμενη συνάδελφο Σενάλοβα, την εισηγήτρια. Θα ακούσουμε τις απόψεις των κυρίων Χάστινγκς, Ρουκ και Νταϊάνι 10 λεπτά ο καθένας. Και μετά θα υπάρξουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Κυρία Σενάλογα όμως πρώτα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν σε αυτήν τη συνάντηση και όσους δέχτηκαν την πρόσκληση αυτή. Το θέμα αυτό για μας είναι ένα κομβικό θέμα και άπτεται της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε έτσι ώστε το σύστημα e-call να διευκολύνει ακόμα περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε ήδη κάνει αρκετές συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό. Νομίζω όμως ότι ορισμένες πλευρές έχουν παραμείνει, θα έλεγα, λίγο θολές. Έτσι λοιπόν, και μετά από την τελευταία μου παρουσίαση, για την εγκατάσταση και την έγκριση τύπου του συστήματος στα οχήματα. Τέθηκαν αρκετά ερωτηματικά, υπήρξαν σχόλια από συναδέλφους, σκιώδεις εισηγητές και γι' αυτό ακριβώς είπαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να οργανώσουμε μια μικρή ακρόαση γύρω από το θέμα. Η σύνθεση νομίζω ε, του hearing αυτού της ε, ακρόασης αυτής είναι αντιπροσωπευτική και χρήσιμη. Θα ακούσουμε τρεις ομιλητές και θα αναφερθούμε στο θέμα της ετοιμότητας των κρατών μελών να αναπτύξουν το σύστημα e-call από το 2015. Θα ακούσουμε επίσης τους συντονιστές, ε, τον συντονιστή κύριο Ρουκ, θα ακούσουμε την παρουσίαση του ελεγκτή προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και κάποια στοιχεία επιπλέον για τον Γαλιλαίο σε σχέση με το e-call. Πρώτα θα ακούσουμε λοιπόν τον ελεγκτή προσωπικών δεδομένων με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί ήδη στο παρελθόν για την προετοιμασία και τροπολογιών, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα βασικό κομμάτι της πρότασης. Χαίρομαι λοιπόν που ο κ. Hastings θα παρουσιάσει τις απόψεις του και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα συμπεράσματά του. Από το 2011 όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το e-call σαν εισηγήτρια για την έκθεση ευθύδιας πρωτοβουλίας και μετά σαν εισηγήτρια για την πρόταση κανονισμού, διαπίστωσα ότι το e-call πρέπει να είναι ένα σύστημα κατεπίγουσας προειδοποίησης που να βασίζεται σε ένα σύστημα το οποίο να δραστηριοποιείται μόνο με το άνοιγμα των airbag. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου συνεχώς και δεν είναι κάτι το οποίο δραστηριοποιείται εκτός οχήματος. Ε, εξεπλάγει λοιπόν από το εύρος των παρατηρήσεων για επιπλέον ιδιωτικές και εμπορικές υπηρεσίες. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ένα δημόσιο σύστημα e-call που βασίζεται στους αριθμούς 112 και 114. Θα ακούσουμε επίσης και την άποψη του κυρίου Ρουκ, ο οποίος γνωρίζει καλά το πρόγραμμα. Ε, θα μας πει τι χρειάζεται να γίνει στα κράτη-μέλη για να αναπτυχθεί σωστά το Ρουκ. Δεν απαιτούνται μόνο συγκεκριμένοι κανόνες, αλλά απαιτούνται και έλεγχοι, δοκιμές κτλ. Βλέπουμε ότι 22 χώρες ε, έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν πιλωτικά προγράμματα σε διαφορετικές συνθήκες που θα ελέγξουν τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες για το e και το στάδιο προετοιμασίας και ετοιμότητας των υποδομών στα πλαίσια της γραμμής 112. Και θα ακούσουμε επίσης ε, και τον κύριο Γιάννη ο οποίος είναι έτοιμος να απαντήσει στα θέματα της ετοιμότητας του Γκαλιλαίου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών e-call. Γιατί όπως λέγει και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία των στοιχείων ανάμεσα στο έγνος και τον Γκαλιλαίο και υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για το στάδιο της προετοιμασίας αυτής και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας, κυρία Σενάλοβα. Εγώ καλωσορίζω τον Πίτερ Χάστινγκ στην ε, συνάντησή μας, είναι τακτικός επισκέπτης. Να τον ευχαριστήσω και εξ ονόματος της Επιτροπής ε, για τις αναλύσεις, τις πολύ χρήσιμες, τις οποίες και λεπτομερείς παίρνουμε για τις εκθέσεις μας. Σας καλωσορίζω και σας δίνω το λόγο λοιπόν κύριε Χάστινγκς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν έρχομαι τόσο συχνά, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για να το κάνω. Πρώτον θα ήθελα να πω ότι ένας από τους βασικούς στόχους της, του ελεγκτή προσωπικών δεδομένων είναι ακριβώς το να παρέχει στοιχεία ε, για θέματα που άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση τις προτάσεις τις οποίες ετοιμάζει να μας τις υποβάλει για να κάνουμε μια μελέτη επιπτώσεων γύρω από τα θέματα της προστασίας των δεδομένων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής σχέση του θέματος με τον τομέα μας. Υπέβαλε τη γνωμοδότησή της στα τέλη Οκτωβρίου να σημειώσω εδώ ότι μια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό γίνεται και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ε, αν και εγώ εκρίνω ότι έπρεπε να έρθω εδώ πρώτα στην δική σας Επιτροπή που είναι η Επιτροπή επί ουσίας. Η συγγήτρια αναφέρθηκε στο θέμα ε, που άπτεται των ε, προσωπικών στοιχείων. Θα πρέπει να τονίσω το εξής εδώ. Το σύστημα e-call τα ιδιωτικά e-call, όπως επίσης και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας γύρω από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και στα οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη έκθεση, θα οδηγήσει στην συλλογή δεδομένων ε, όταν κινούνται τα οχήματα, όταν κινούνται οι οδηγοί των οχημάτων θα χρησιμοποιηθεί ο λεγόμενος γεωεντοπισμός και γενικότερα άλλα ευαίσθητα θέματα. Δηλαδή το σχέδιο σχεδιάστηκε, το σχέδιο μάλλον προετοιμάστηκε για να βοηθήσει σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τμήμα υποδομών το οποίο θα οδηγήσει στην, στον γεωεντοπισμό ή περνάει μέσα από το γεωεντοπισμό. Οπότε εδώ αυτόματα υπάρχει μια υποχρεωτική απώλεια ιδιωτικών στοιχείων είτε είναι τμήμα ε, της ιδιωτικής πλατφόρμας e-call, είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιατρικές υπηρεσίες, νοσοκομιακές υπηρεσίες κτλ. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να αναλύσουμε την κατάσταση αυτή και φτάσαμε στα πρώτα συμπεράσματα τα οποία λέγουν ότι σε σχέση με αυτούς ε, που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα και τίθεται εδώ το θέμα, τίθεται ήδη δηλαδή γιατί ήδη χρησιμοποιείται το σύστημα σε εθελοντική βάση. Η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία υπάρχει και η εθνική νομοθεσία θα ισχύσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και γι' αυτό λοιπόν θα υπάρξουν κανόνες οι οποίοι θα αφορούν το μελλοντικό αυτό ε, σύστημα. Η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντική. Περνάει από μια εθελοντική ε, ε, κατασκευή e 112 σε ένα υποχρεωτικό σύστημα 112, αριθμός κλήσης δηλαδή πρώτων βοηθειών. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα παρέχουν ε, την, το χαρακτηριστικό αυτό, την εφαρμογή αυτή, σε μια ασφαλή και σεβόμενη τα ιδιωτικά στοιχεία βάση. Δηλαδή μιλάμε για ιδιωτικά στοιχεία από τη στιγμή που σχεδιάζεται το προϊόν, το αυτοκίνητο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως δείχνει η γνωμοδότηση, υπάρχουν κάποια θέματα που είναι σε εκκρεμότητα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε εδώ ότι κάθε φορά που ο κοινοτικός νομοθέτης ε, που ασχολείται με τα θέματα του άρθρου 114, δηλαδή την εσωτερική αγορά και ασχολείται με πλευρές που άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ένα τμήμα της νομοθετικής αυτής της διαδικασίας προβλέπει την δημιουργία ρητρών ασφαλείας, αν θέλετε, έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα της κοινότητας. Και ναι μεν χρησιμοποιείται το 114 σαν νομική βάση, αλλά πρέπει όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα άρθρα 7 και 8 της χάρτας, όπως επίσης και του άρθρου 60. Αυτό τι σημαίνει. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Αν αυτές οι συμπληρωματικές ρήτρες ασφαλείας δεν είναι κατάλληλες πλήρως. Η μελλοντική νομοθεσία θα αμφισβητηθεί ως ασύμβατη με τις συνθήκες. Ή οι χρήστες αυτών των ιδιωτικών ε, μεθόδων αν θέλετε θα έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολα θέματα τα οποία δεν μπορούν να το κάνουν αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες νομικές ρυθμίσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα δεν είναι να είναι κανείς ριζοσπάστης, αλλά να διασφαλίσει ότι η αγορά θα παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω αυτής της εξαιρετικής υποδομής. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία γραπτά που αναφέρονται σε αυτές τις επιπλέον διαστάσεις. Δεν θα επαναλάβω εδώ όλες τις λεπτομέρειες των γνωμοδοτήσεων, αλλά το βασικό στοιχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η πρόταση ως έχει συγκεντρώνεται μόνον σε δημόσια χρήση του e-call αριθμός κλήσης 112. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ο ιδιωτικός τομέας εδώ δεν φύγεται ουσιαστικά. Το βασικό θέμα λοιπόν που τίθεται το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ε, μια συγκεκριμένη συνένεση έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες αυτές και από τον ιδιωτικό τομέα. Ε, και σε ποιο βαθμό ο ιδιωτικός τομέας έχει τη δυνατότητα της γεωπαρακολούθησης, γεωεντοπισμού κτλ. Αυτά είναι θέματα που δεν έχουν τεθεί όπως είπαμε ακόμα. Η πρόταση ε, ξεπερνά αν θέλετε κάποια όρια, αυτή είναι η γνώμη μας και προσπαθεί να ορίσει ακριβώς τις ρήτρες προστασίας που απαιτούν και προϋποθέτουν τη συνένεση των Χριστών. Το κείμενο λοιπόν απαιτεί να υπάρξει σωστή ενημέρωση για να υπάρξει ε, σωστή και τεκμηριωμένη συνένεση, αφορά και άλλες υπηρεσίες, ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν να ασχοληθεί κανείς με την ε, εναλλακτική πρόταση ή την αρχικά καθορισμένη κατάσταση στη λειτουργία του συστήματος. και να μιλήσω με λίγες περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα αντιμετωπιστούν μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων και κάποια άλλα μη σημαντικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αναφερθεί καθόλου στην οδηγία έτσι όπως προτείνεται, στον κανονισμό τον οποίο προτείνεται. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα επιπλέον και σε σχέση με την ενημέρωση για να υπάρχει τεκμηριωμένη συνένεση και αν η ενημέρωση, οι πληροφορίες παρέχεται ε, μέσω εγγράφων σαν παράδειγμα που είναι μέσα στο αυτοκίνητο ε, το οποίο σπανίως διαβάζουν οι χρήστες των αυτοκινήτων οι οδηγοί τότε φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξει σωστή ενημέρωση. Υπάρχει λοιπόν λόγος έτσι ώστε όταν αρχίζει να λειτουργεί το σύστημα δεν αποφασίζει κανείς εκείνη τη στιγμή και μιλάω για το κανονικό GPS ε, για θέματα όπως επιλογή δρόμων με διόδια ε, και κτλ ή χωρίς διόδια, αλλά να σου λέει το σύστημα ότι παρακολουθήσε, εντοπίζεσαι ηλεκτρονικά συνεχώς, το δέχεσαι ή όχι. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μία νομική υποχρέωση, όπου οι συνέπειες, ε, τα προερχόμενα στοιχεία αν θέλετε, της χρήσης του συστήματος θα πρέπει να κρυθούν αποδεκτά ή όχι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια επιμέρους στοιχεία τα οποία θα ήθελα να σας μεταφέρω, κάποια από αυτά τα ανέφερα ήδη. Σαν παράδειγμα την ανάγκη ε, απαγόρευσης της συνεχούς παρακολούθησης ε, για εμπορικούς λόγους, κάποια βασικά στοιχεία για τους τρόπους και τις μεθόδους και τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων, η διασφάλιση ακριβώς της ασφάλειας της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων, εδώ τίθεται θέμα της τεχνολογίας η οποία χρησιμοποιείται και τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ε, η ενημέρωση, το δελτίο, το ενημερωτικό σε θέματα ασφαλείας οι τρόποι με τους οποίους θα απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων εφόσον υπάρχει έλλειψη συνένεσης. Ήδη κάποια πρώτα στοιχεία έχουν εφαρμοθεί σε διάφορες χώρες με κάποιες μικρές διαφορές σεβόμενοι την εσωτερική αγορά. Πρέπει αυτό να το κατανοήσει ο χρήστης, να γίνεται αναφορά σε αυτό το στοιχείο και υπάρχουν και δύο στρατηγικές επιλογές εδώ οι οποίες θα πρέπει να απασχολήσουν. Γιατί εσείς θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες και από το θέμα αυτό. Τα επιπλέον βήματα θα πρέπει να είναι σε επίπεδο mainline, δηλαδή κυρίαρχο. Και από την άλλη δημιουργεί κανείς ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ένα κίνητο, όχι μόνο στην αιτιολογική σκέψη αλλά και στις ε, ρήτρε απόφασης που απαιτούν από τους εθνικούς νομοθέτες να, καθοδηγούν και αυτό το έχει ζητήσει και η ομάδα του άρθρου 29. Κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν και προς τη βιομηχανία πριν την παραγωγή των συστημάτων. Ήδη έχουν ζητήσει πληροφορίες ε, οι βιομηχανικοί κύκλοι. Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, περισσότερες πληροφορίες. Το να αγνοήσουμε το αίτημα αυτό δεν θα ήταν καλό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είναι σε εκκρεμότητα κατά κύριο λόγο και μετά να αναφερθούμε στις επιπλέον ε, μορφές ενημέρωσης, πληροφόρησης ε, των εμπλεκομένων. Έτσι ώστε αυτό το ζωτικό αν θέλετε ε, εργαλείο να, μην, να γίνει εύκολα ή ευκολότερα κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις παρουσίασή σας και για την πολύ ρεαλιστική παρουσίασή σας σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το βασικό θέμα που θα συζητήσουμε. Αυτό λοιπόν ε, το λέω και ως κοιόδης, όχι μόνο ως πρόεδρος της Επιτροπής. Μάλιστα, θα συγκεντρώσουμε λοιπόν όλες τις ερωτήσεις μαζί στο τέλος και ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες επικαλύψεις Με ιδιαίτερη χαρά μου λοιπόν καλωσορίζω τον Αντιρούπ να μας μιλήσει. Είναι σημαντικά αυτά για να καταλάβουμε πόσο ε, έχει, που έχει φτάσει το e-call και με μια εφαρμογή που νομίζεται πρόγραμμα Hero Φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ε, για να θυμόμαστε λοιπόν τέτοια project. Το Hero Project λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνει το λόγο να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα αυτό. Πρόκειται αυτή την, αυτά τα θέματα θέλω να καλύψω σε ό,τι αφορά τις προπτικές του Hero Project, ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι, τεχνικοί τομείς που καλύπτονται Πολύ σημαντικό αυτό για τη συζήτηση που ήδη έχει λάβει η χώρα. Το χρονοδιάγραμμα που βρισκόμαστε στην παρούσα φάση και μια ενημέρωση σε ό,τι αφορά το καθεστώς των 15 πιλωτικών ιστοσελίδων ε, που διαθέτουμε και κάποιες παρατηρήσεις από τα τρία χρόνια εμπειρίας μας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή δηλαδή και τη χρήση του e-call. Για τα μέλη εκείνα που δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς λειτουργεί το e-call, μία πολύ σύντομη παρουσίαση με απλούς όρους. Η τεχνολογία κινητών τηλεφώνων που έχει ενσωματωθεί στα οχήματα ε, με πρόσβαση στην ε, κινητή τηλεφωνία και χρησιμοποιεί σήματα GNSS και έτσι τίθεται σε εφαρμογή τα αυτόματα ή τα χειροκίνητα και αποστέλει μία μικρή ομάδα δεδομένων σε ένα σημείο κόμβο που ε, κρυπτογραφεί και επιτρέπει την επικοινωνία με το όχημα. Αυτό το είναι το e με πολύ, με πολύ απλά λόγια όλες ε, οι κλήσεις γίνονται μέσω του δικτύου 112. Δεν υπάρχουν ιδιωτικέ κλήσεις, δεν ε, εμπλέκονται τρίτη φορείς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτές λοιπόν είναι οι προπτικές σε ό,τι αφορά το project. Ξεκινήσαμε τον ε, Ιανουάριο του 2011 και θα ολοκληρώσουμε το έργο μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Έχουμε 15 πληθυντικά τοποθεσίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, συνεταιριζόμενες χώρες. 8 εκατομμύρια ευρώ έχουμε για τα δύο project, χρηματοδότηση, 15% δηλαδή ποσοστό. Άρα υπάρχει μια δέσμευση από, τη, από τους εταίρους. Έχουμε 82 εταίρους συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των πληθυκών τοποθεσιών. Μετά την εισαγωγή του δεύτερου Project Hero. Μας προσέγγισαν αρκετά κράτη-μέλη και συνδεόμενες χώρες που αναγνώρισαν ότι το e-call χρειαζόταν και ζήτησαν την ερωγή μας για να καταλάβουν ακριβώς τι είναι το e-call. Προκειμένου να μπορέσει το οικοδόμημά του σε ό,τι αφορά τις ε, κινητή τηλεφωνία να ενημερωθεί, να ανα βαθμιστεί και η Ρωσία, να σας πω ότι έχει ένα πολύ παρόμοιο σύστημα και είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία. Δυστυχώς το Ισραήλ δεν είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε το κάνουμε. Πάντως η κατάσταση αλλάζει. Ε, ήδη την προηγούμενη εβδομάδα η Ιρλανδία συμμετέχει ως συνδεδεμένη χώρα και ζήτησε ε, την βοήθεια για να αντιληφθεί πώς πρέπει να διαμορφωθεί το δίκτυο τηλεφωνίας για να υποστηρίξει το e-call. Αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας τώρα είναι η στόχη του προγράμματος HERO. Αρχικά είχε μια θεωρητική προσέγγιση στο μέσον του Hero 1 όταν εγώ ασχολήθηκα με το πρόγραμμα ε, φρόντισα οι στόχοι να γίνουν πιο συγκεκριμένοι. Πρέπει να, ε, ε, να δούμε πώς αυτό το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, πώς μπορεί να ενισχυθούν οι επενδύσεις στο e-call και γενικά να υπάρξει μια μεγαλύτερη υιοθέτηση του συστήματος. Αυτό το προωθήσαμε μέσω των συνδεδεμένων περιοχών. Τεχνικά ζητήματα Ήδη αναφέρθηκαν τα διαφορετικά είδη e-call που υπάρχουν. Ο κύριος στόχος ο δικός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο e-call βασιζόμενο στο ε, αριθμό κλήσης 112 για τα οχήματα τύπου M1 και N1, δηλαδή τα ιδιωτική χρήσης ε, οχήματα μέχρι 5 θέσεις και μέχρι ε, τόνους ε, φορτίο. Όμως, προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπέρα. Εξετάζουμε τη δυνατότητα τη αγωγή του e-call για, σε φορτηγά και κυρίως εκείνα που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. Το εξετάζουμε επίσης για τα δίκυκλα που είναι ιδιαίτερα ε, κινδυνεύουν στους, στους, στους δρόμους της Ευρώπης. Εξετάζουμε επίσης την χρήση πολλών συστημάτων πλοήγησης, καθώς επίσης και τη δρομολόγηση της κλίσης 112, ε, έτσι ώστε να καταλήγει στο σωστό κέντρο. Αν εναλλακτικές συσκευές με βάση τον αριθμό των αυτοκινήτων που, είναι, που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, διαπιστώνουμε ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια, πολύ, πολύς χρόνος μάλλον, για να γενικευτεί η χρήση του, μιας και ο κανονισμός αναφέρεται μόνο στα νέα οχήματα που θα κυκλοφορήσουν μετά το 2015. Οι συνάδελφοί μου στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ε, έχουν επισημάνει ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα που σχετίζεται με την ανανέωση του στόλου στις χώρες τους, έτσι ώστε τελικά όλοι οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους το e-call. Μετά, Υπάρχει το ζήτημα της πιστοποίησης των οχημάτων που ήδη βρίσκονται στην κυκλοφορία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι από τη στιγμή που εισάγεται ένα σύστημα e-call σε ένα όχημα θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του. Θα πρέπει να μην υπάρχουν λανθασμένες κλήσεις και όταν γίνεται μια κλήση e-call αυτή να έχει γίνει για το σωστό λόγο. Όταν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Δημιουργούμε πρότυπα για τον έλεγχο. Βλέπετε εδώ το χρονοδιάγραμμα και που βρισκόμαστε. Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μέρος του προγράμματος και ετοιμάζουμε την έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος του Hero 1 που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Στην αριστερή πλευρά. Η Κροατία ολοκλήρωσε τις δοκιμές και η Κροατία είναι πλήρως έτοιμη να υποδεχθεί και να ε, υποστηρίξει το πρόγραμμα E-Call. Τσεχία. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και στη χώρα αυτή μπορεί να εφαρμοστεί το E-Call. Φινλανδία. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος συνεργασία με τη Ρωσία και αναμένει το σύστημα PSAP, το οποίο θα αρχίσει να χρησιμοποιείται από το 2015. Έχουν γίνει οι ε, προσκλήσεις ε, για δημοπρασία, για δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια αυτών του εξοπλισμού. Γερμανία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αλλά εδώ είναι πιο περίπλοκη η κατάσταση. Έχει δημιουργηθεί ένα ε, μοντέλο σε μία περιοχή της ε, Γερμανίας που θα μπορούσε να γενικευτεί και στις υπόλοιπες. Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε εδώ είναι περίπλοκα και έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες αυτή η χώρα φέτος και πέρυσι. Καταφέραμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικά για την Ελλάδα έξι μήνες παράταση. Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται τώρα και με την εξάμεινη παράταση θα καταφέρουν να είναι έτοιμοι στην ώρα τους. Ιταλία ολοκλήρωσε τον έλεγχο και έχει ένα σύστημα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Ιταλία. Υπάρχει παράλληλα μια διαδικασία αναθεώρησης του συστήματος του 112 στην Ιταλία. Ρουμανία Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, είναι πλήρως έτοιμη να εφαρμόσει το σύστημα παντού. Σουηδία ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και πάλι εδώ αναμένουν μια πολιτική απόφαση. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν με το χειρού 1 και ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουάριο χείρο 2. Βρισκόμαστε περίπου στο τέλος της πρώτης χρονιάς. Εδώ έχουμε αξιοποιήσει τα διδάγματα από το πρώτο πρόγραμμα και έχουμε τροποποιήσει κάπως την προσέγγιση μας. Όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο χείρο 2 πρέπει να παράσχουν ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου θα γίνει ο έλεγχος. Θα σας εξηγήσω γιατί αργότερα. Ωστόσο, πολλά κράτη-μέλη έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για το φόρτο που θα δημιουργηθεί στο κέντρο που απαντά τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίω σε περιπτώσεις που γίνονται κλήσεις χωρίς να ε, ε, μιλήσει ο καλόν. Ε, το Βέλγιο και η Ισπανία εξετάζει μια τεχνολογία που θα μπορούσε να κάνει screening, να ελέγχει αυτές τις κλήσεις για να δει αν είναι πραγματικές. Το βελγικό σύστημα το έχει αναπτύξει μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά έχει αγοράσει τα δικαιώματα χρήσης του το, η βελγική κυβέρνηση. Η Ισπανία ε, σκέφτεται, προτιμά μια δημόσια λύση. Η Δανία είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα πρόσβασης στο PSAP, αλλά είναι η μόνη χώρα στην οποία θα εξεταστεί η χρήση μιας ανενεργούς ε, κάρτας SIM. Αυτές οι ενεργές κάρτες SIM, κατά την άποψή μου, είναι η το θεμέλιο της ε, δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος e γιατί δεν ε, παρακολουθούν το χρήστη τους, απλώς ενεργοποιούνται όταν χρειάζεται. Λουξεμβούργο. Εξετάζουν και εκείνοι το σύστημα πανευρωπαϊκού e-call, Ισπανία επίσης και η Τουρκία. Δεν σας αναφερθώ τώρα στην τυποποίηση γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και έρχομαι στις παρατηρήσεις μου από τα δύο αυτά προγράμματα. Τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο HERO αναμένουν την πρόοδο στις νομοθετικές ε, παρεμβάσεις και ζητούν μεγαλύτερη σαφήνεια. Η διατύπωση της ε, φόρμας συνένεσης δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη και θα πρέπει να βελτιωθεί. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι εξαιρετική σημασία για το πανευρωπαϊκό Το GSMA υποστηρίζει ένα πανευρωπαϊκό e-call και υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασία. Αλλά η κατάσταση είναι διαφορετική από, μέλος, από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα αυτό. να... Υπάρχουν πολλά συναρμόδια υπουργεία, μέχρι και πέντε σε κάποιε χώρε. Θα αλλάξουν οι διαδικασίες λειτουργίας εξαιτίας του e και τέλος, είναι σημαντικό, να σκεφτούμε πώς θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτό στους πολίτες της Ευρώπης. Αυτά από την πλευρά μου κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις ε, για το θέμα αυτό αργότερα, σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά τεχνολογίες. Όπως είπατε, χρησιμοποιείται η Αν η ενυπνώση SIM. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποίησατε. Η κυρία Διάννη. επειδή βασικά ε, βασιζόμαστε στο e-call στη γεωγραφική τοποθέτηση. Και θα μας μιλήσετε λοιπόν για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να σας εξηγήσω το θέμα της ε, τοποθεσίας ε, σε ό,τι αφορά το e-call και το θέμα της ε, πλοήγησης μέσω δορυφόρου. Έγνος και Γαλιλαίος. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είμαι μηχανικός αεροδιαστήματος. Ξέρω ότι σε κάποιες περιστάσεις ε, μιλάμε για και χρησιμοποιούμε όρους, ακρονίμια, έτσι, φυσικής. Θα προσπαθήσω όμως στη δική μου παρουσίαση να τα αποφύγω αυτά. Θα ζητώ συγγνώμη και των προτέρων αν σε κάποιες περιπτώσεις ε, χρησιμοποιώ κάποια περίεργα ακρονίμια. Καταρχάς, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω γιατί η ακριβής και αξιόπιστη τοποθέτηση σημαίνει με ζωές που σώζονται για να βρούμε την ακριβή ε, τοποθεσία του e-call. Ε, αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες ε, επίγουσας ανάγκης μπορούν να βρουν την τοποθεσία του ατόμου που χρειάζεται βοήθεια και επίσης αυτό μπορεί να βελτιώσει δραστικά το χρόνο παρέμβαση σε περίπτωση σιωπηρών κλήσεων και σε περίπτωση προστή που δεν υπάρχει διαθέσιμη φωνή και ε, κάποιος ε, θόρυβος, μπορούμε με ακρίβεια να υπολογίσουμε την υποθεσία του e-call. Τι είναι λοιπόν, πώς ε, συμβάλλουν τα προγράμματα αυτά και η Ευρώπη στην πλοήγηση αυτή. Το έκνος είναι ένα πρόγραμμα βελτίωσης ε, του GPS, το σύστημα που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα, στα κινητά μας τηλέφωνα. Βελτιώνει την εγκυρότητα και την ακρίβεια του GPS στο έγνος και δίνει καλύτερο, καλύτερη αξιοπιστία, και καλύτερη τοποθεσία σε ό,τι αφορά το σήμα. Είναι λειτουργικό από το 2009 και η ανοιχτή υπηρεσία είναι δωρεάν. Το σύστημα Γαλιλαίο αποτελεί το παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης, το οποίο είναι Made in EU και είναι απόλυτα ασύμβατο με το GPS. Το Γαλιλαίο λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπρόσθετο σύστημα δορυφορικό σε συνδυασμό με το GPS. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι πλήρης η εφαρμογή. Είναι βελτιώνει το σύστημα αυτό. Η αρχική λειτουργική η υπηρεσία του Γαλιλαίου προβλέπεται από το τέλος του 2014 και η αρνητική υπηρεσία επίσης είναι δωρεάν. Να σας δώσω τώρα κάποια παραδείγματα το πώς το έγνος και το Γαλιλαίο μπορούν να βελτιώσουν την τοποθεσία e-call. Καταρχάς, ας σκεφτούμε μία απόμακρη περιοχή στην Ήπεθρο. Φυσικά η ακρίβεια της τοποθεσίας είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αν μπορούμε να διακρίνουμε κατά πόσον το ατύχημα έγινε στο δικό δικτύο ή εκτός ε, οδικού δικτύου, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι ο δίκτυπος σε ό,τι αφορά την ε, παρέμβαση, σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα του ατυχήματο. Ας κοιτάξουμε και το αστικό περιβάλλον. Στο αστικό περιβάλλον υπάρχουν τα επωνομαζόμενα φαράγγια, αστικά φαράγγια, όπου υπάρχει για παράδειγμα παρεμπόδιση του σήματος. Άρα μπορεί να υπάρχει καλή δορυφορική επαφή ε, συνδυάζοντα ε, το GPS με τον καλλιλέο. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ακρίβεια και την διαθεσιμότητα του σήματος και της τοποθεσίας δηλαδή του ατυχήματο για να απαντήσω στο ερώτημα του κατά πόσον το σύστημα, αυτή η υποδομή του της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λειτουργικά. Σε ό,τι αφορά το έκνο, σας είπα, είναι λειτουργικό από το 2009 και μετά. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις ανακοινώσεις του τύπου του 1 Οκτωβρίου 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώνει την ε, λειτουργικότητα των ε, υπηρεσιών έγνος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Enterprise έκανε και κατευθείαν μία μελέτη το 2010-2011 για να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα του έγνος για, τα, για την εφαρμογή. Τα αποτελέσματα και τα πορίσματα παρουσιάστηκαν σε διάφορες περιστάσεις και υπήρξε γενικά ενημέρωση για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά το Γαλιλαίο τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει για να φέρουμε τον Γαλιλαίο. Έχουμε πλέον εκτοξεύσει τέσσερις δορυφόρους που ήδη συμμετέχουν στη λειτουργική οικογένεια δορυφόρων από τον Οκτώβριο του 2012. Όλες οι βιομηχανικές συμβάσεις ε, που χρειάζονται για τους δορυφόρους έχουν υπογραφεί και οι πρώτες υπηρεσίες ε, προγραμματίζονται για τα τέλη του 2014. Τον Μάρτιο του 2013 Ζήσαμε μια συναρπαστική στιγμή, γιατί το πρόγραμμα Γαλιλαίο άρχισε να εκπέμπει το σήμα πλοήγησης σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, λοιπόν, την ίδια ημέρα, πολλοί ειδικοί GNSS, αυτοί δηλαδή που κατασκεύασαν τις συσκευές, και επιστήμονες υπολόγισαν τις πρώτες θέσεις βάσει του Γαλιλαίου, υπολόγισαν την είναι εξαιρετικό το σήμα και πραγματικά πρωτοποριακό σε ό,τι αφορά τη τεχνολογία τη δορυφορική. Για να απαντήσουμε τώρα το ερώτημα κατά πόσον τα συστήματα αυτά, κατά πόσον τα υποδομές αυτές είναι ε, χρήσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η βελτίωση του δορυφορικού σήματος που αποτελεί τμήμα στο οποίο υπάγεται το έγνος αποτελεί μία, ένα κοινό τόπο σε ό,τι αφορά τις συσκευές λήψης σήματος, σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα πολύ συστηματικά, καθίστανται σημεία αναφοράς. Ε, έχουμε ήδη ε, smartphones και έχει γίνει μία ανάλυση στο GSA βάσει ανεξάρτητων πηγών, Genius Word, μία από τις πιο έγκυρες ε, εταιρείε και υπολογίσαμε λοιπόν ότι φέτος ήδη το 40% των εκπομπών λήψης για την χρήση σε αυτοκίνητα είναι συμβατή, συμβατό με το Γαλιλαίο και ότι 60% έχουν δυνατότητα χρήσης του έγνος. Αυτό βελτιώνει κατά 10% τα μοντέλα ε, συσκευών λήψης σήματος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πραγματικά διατίθενται αυτές οι υποδομές. Για να διευκολύνουμε όμως αυτή τη διαδικασία, ήδη φέτος το καλοκαίρι, μετά από την πρόταση του σχετικού κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δώσαμε τη δυνατότητα για τους κατασκευαστές ε, ε, συσκευών λήψης. και τον τσιπ. η ειδικοί μας ε, και που έχουν λάβει την κατασκευή του Γαλιλαίου να ελέγξουν λοιπόν την συμπατότητα με τον Γαλιλαίο. Οι πιο πολλοί κατασκευαστές λοιπόν από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική, στη φάση, καθότι είχε ήδη ολοκληρωθεί η φάση ελέγχου, θεωρούμε λοιπόν ότι θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν από το Ιανουάριο. Αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί ένα καλό τρόπο εφαρμογής των ε, εμπειριών μας. Ένα άλλο βήμα είναι, ήταν η διαβούλευση με τον βιομηχανικό κλάδο των, ε, δηλαδή των συσκευών αυτών, των αποδεκτών και των τσίπ. Μας ζήτησαν την ε, υποστήριξή μας για να ελέγξουν τις ίδιες τις συσκευές. Τους δώσαμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία σε συνεργασία με το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήδη έχει δημοσιευθεί η δήλωση ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τους κατασκευαστές των συσκευών αυτών, προκειμένου να ελεγχθεί η συμβατότητα με το Γαλιλαίο σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο. Ας πράσω στα βασικά μηνύματα στα οποία ήθελα να σας δώσω. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι το e-call ωφελείται πολύ σημαντικά από τη διαθεσιμότητα των νέων ικανοτήτων, των νέων δυνατοτήτων GNSS σε ό,τι αφορά τώρα την ευρωπαϊκή συμβολή, το έγνος και τον Γαλιλαίο. Το έγνος είναι βασικά για την Ήπεθρο, το Γαλιλαίο για τις αστικές περιφέρειες. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι θα ωφεληθεί έμεσα και το και το e Αυτές οι δυνατότητες λοιπόν είναι κάτι το κοινό πλέον στην αγορά, αλλά θα πρέπει να τα ζητούν συγκεκριμένα οι καταναλωτές. Θεωρούμε ότι χρειάζεται να ενταχθεί μια δυνατότητα βελτίωσης και στο μέλλον των συστημάτων e-call για να συμπεριλαμβάνουν και τα νέα GNSS. Προκειμένου να βελτιωθεί και η σχέση κόστους και απόδοσης για το κάθε όχημα. Προσφέραμε επίσης ε, την υποστήριξή μας για να διευκολυθεί η φάση ελέγχου και αυτό σε συνεργασία με το Project Hero το οποίο παρουσίασαν οι συνάδελφοι πριν από λίγο προκειμένου να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και τις δικές τους συστάσεις αλλά και τις δικές τους εμπειρίες και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα περισσότερο. No, you Ήσασταν σαφεστάτη και επανειλημμένα έχουμε ακούσει πληροφορίες και είχαμε σωστή ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα Γαλιλαίου γιατί είμαστε υπεύθυνοι επί της ουσίας. Η εισηγήτρια θα ήθελε να θέσει ερωτήσεις. Κυρία Ρούλε, ο κύριος Σοσβάμπ, θέλετε να ξεκινήσετε τις ερωτήσεις κυρία Σενάλοβα. Αφού μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις θα ζητήσουμε από τους ομιλητές μας να δώσουν τις απαντήσεις. Και μπορούν να θέσουν και ερωτήσεις ο ένας τον άλλο αν θέλουν, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει επίσης και ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν κάποιος κύριος ε, προηγουμένως εδώ, αλλά αν θέλουν το λόγο θα τους τον δώσουμε. Να ξεκινήσει η κυρία Σενάλογα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Έχω λίγες ερωτήσεις και ένα σχόλιο να κάνω. γνωρίζουμε τώρα ποια είναι η κατάσταση και στις συνδεόμενες χώρες και στις ε, ε, χώρες μέλη. Αλλά τι γίνεται με τις χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πιλωτικό χέρο. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση την οποία θα είχα να θέσω. Η δεύτερη είναι ότι ζητάμε την ανάπταξη του συστήματος από, τις, ε, από την 1η Οκτωβρίου του 2015. Ορισμένες χώρες όμως έχουν πολλές αμφιβολίες αν κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό. Πιστεύετε ότι υπάρχει δυνατότητα τήρησης του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά τον κύριο Χάστινγκς. Φυσικά και θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι υπάρχει μια βασική διαφορά από ένα δημόσιο e-call που βασίζεται στην κλίση του 112 που αυτός είναι ο στόχος του συγκεκριμένου κανονισμού και από την άλλη στην ιδιωτική ε, εμπορική χρήση του συστήματος που είναι εκτός ε, του πεδίου της συγκεκριμένης αυτής ρύθμισης. Φυσικά και όλα τα σχόλια τα οποία αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία μας παρουσίασε και μας έστειλε ο κύριος Χάστινγκ τον μήνα Οκτώβριο έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χάστινγκς και νομίζω ότι καλύπτονται εν από κάποιες ε, τροπολογίες πολλών συναδέλφων και του συναδέλφου εισηγητή στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Έχω καταθέσει και εγώ η ιδία ε, σαν εισηγήτρια κάποιες τροπολογίες, αλλά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει μάλλον μια κάποια συμφωνία η διεύρυνση ε, του πεδίου του κανονισμού σε υπηρεσίες παρεχόμενες από τρίτους. Το θέμα της ανοιχτής πλατφόρμας όπως επίσης και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία βρίσκονται εκτός του πεδίου της προτινόμενης νομικής ρύθμισης. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο για την ανοιχτή πλατφόρμα σχετικά με την τροπολογία 9 Εδώ το θέμα απαιτεί κάποιες επιμέρους νομικές ρυθμίσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έρθει σε επαφή και να διαβουλευτεί με όλους τους αξιολογητές τις χώρες που αξιολογούν δηλαδή έτσι ώστε να υπάρξει ε, ε, υποβολή μιας νομοθετικής πρότασης αν αυτή η πράγματι χρειάζεται. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι το πολύ συγκεκριμένο και αυτή η πρόταση θα πρέπει φυσικά να σέβεται και τα προσωπικά δεδομένα. Να σχολιάσω επίσης και την τροπολογία υπαριθμών 6 εδώ λέγω ότι κάθε συμπληρωματική υπηρεσία θα πρέπει να έχει γίνει αντικείμενο σχεδιασμού με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην απασχολεί τον οδηγό και να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας, οδήγησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και επαναλαμβάνω, οι υπηρεσίες αυτές παραμένουν εθαλοντικού τύπου. Και έρχομαι εδώ στο θέμα του ιδιωτικού e-call ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει εάν θα δεχθεί να υπάρχουν συμπληρωματικές εμπορικές υπηρεσίες πέραν της συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας του e-call. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Τα ιδιωτικά συστήματα ήδη προσφέρονται από την αγορά καλύπτονται από συμβατικές ρυθμίσεις ανάμεσα στον κατασκευαστή από τη μία και τον καταναλωτή από την άλλη. Και έρχομαι εδώ σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο έθεσε ο Ροκ και είναι κάτι το οποίο έπρεπε να αναφέρω και εγώ. Είναι η λεγόμενη κάρτα SIM ενυπνώση, στην οποία βασίζεται ε, το ε, e-call δεν είναι εγγεγραμμένη στο δίκτυο και δεν επιτρέπει την παρακολούθηση από τρίτους του οχήματος. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα το οποίο πρέπει να ξεχωρίσουμε και είναι κάτι που ξεχωρίζει το σύστημά μας. Ευχαριστώ. κύριε Σβάμπ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα και εγώ με πάρα πολύ προσοχή τις ε, παρεμβάσεις αυτές και δεν ήθελα να επαναλάβω το οτιδήποτε. Θα ήθελα αυτά που είπε η κυρία Σενάλοβα στο τέλος ε, να τα θέσω ε, ως ερώτηση για τον υποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς πώς το τοποθετηθήκατε. Άρα, κύρια Χάστινγκς, πιστεύετε ότι είναι προβληματικό να υπάρξει μια ρύθμιση για να μπορεί μέσω κάρτας μία κλίση ε, ενός ε, όπου δεν υπάρχει, όπου υπάρχει ένα τύχημα σε αυτοκίνητο και σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η παρέμβαση του airbag, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι δεσμευτικό και τι όχι. Um, any other Κανείς άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Έχω και εγώ κάποια θέματα να σας θέσω. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον κύριο Ρουκ, προς τον κύριο Ρουκ. Αναφερθήκατε σε κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Ίσως αυτό βέβαια να μην είναι ακριβώς της αρμοδιότητας της, αλλά υπάρχουν ανεπίλητα ζητήματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία έχω μιλήσει με κάποιους αξιωματούχους και ε, ε, αμφιβάλλουν για τη σχέση κόστους-οφέλους του συστήματος. Δεν είναι όλοι πεπισμένοι λοιπόν. Και ρωτώ, όπου έχει εφαρμοστεί πιλωτικά αυτό το σύστημα, μήπως έχουμε συλλέξει στοιχεία Μήπω έχουμε στη διάθεση μα λοιπόν στοιχεία για να προχωρήσουμε. Για την παρουσία τη κυρία Διάννη θα ήθελα να ρωτήσω. Σα καλύπτουν οι υφιστάμενε διατάξεις γιατί διάφορα ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη πει ότι θα έπρεπε το σύστημα Γαλιλαίο να συμπεριληφθεί αλλά οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι ακόμα διαθέσιμες και άρα το χρονοδιάγραμμα είναι μη ρεαλιστικό για να αξιοποιηθεί το σύστημα Γαλιλαίο. Η εντύπωση που μου δόθηκε από την ε, παρουσίασή σας είναι ότι συμφωνείτε εσείς με αυτό, αλλά θα ήθελα να μου το εξηγήσετε καλύτερα. Τώρα, για τον κύριο Χάστινγκς. θίξατε στο τέλος. Τι γεγονό ότι θα πρέπει να είναι πιο σαφείς οι κατευθυντήριες οδηγίες που θα δοθούν για όλα τα συστήματα ε, παρακολούθησης, γεωπαρακολούθησης που ήδη ε, χρησιμοποιούνται. Το e-call είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα, πολύ περιορισμένο. Πρόκειται για ένα σύστημα δημόσιας χρήσης, εντελώς ε, ανώνυμο γιατί αυτό το, τα δεδομένα τα οποία μεταδίδονται δεν αναφέρονται σε κανένα άτομο, σε κανένα πρόσωπο συγκεκριμένα. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του οδηγού. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει πρόβλημα προσθέσεις προσωπικών δεδομένων. Αντιλαμβάνομαι το ζήτημα που ανακύπτει όταν μιλάμε για υπηρεσίε προστιθέμενες αξίες, για τις εμπορικές χρήσεις αλλά εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία αναφέρεται στο όχημα και δίνει τη δυνατότητα ε, οι αερόσακοι να ξεκινούν μια διαδικασία ε, μετάδοσης ενός ανώνυμου συστήματος, ε, Και είχαμε μια παρουσίαση του πιλωτικού προγράμματος από την Τσεχία και είδαμε ότι τα σήματα που μεταδίδει το όχημα είναι αρκετές φορές περίπλοκα γιατί μας δίνουν για παράδειγμα τον αριθμό των αερόσοκων που ε, άνοιξαν, που ίσως μας δώσει μια αίσθηση του σοβαρότητας του ατυχήματος κτλ. Αλλά υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα για όλα αυτά τα συστήματα εντός οχήματος και το GPS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για γεωπαρακολούθηση. Όλα αυτά τα συστήματα γεωπαρακολούθησης θέτουν στο χρήστη τους κάθε φορά το ερώτημα αν συμφωνεί με συγκεκριμένους όρους χρήσης. Υπάρχουν λοιπόν ευρύτερα θέματα, τα οποία δεν έχουν τόσο σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, αλλά για παράδειγμα με την μετάδοση στοιχείων τεχνικής φύσεως γιατί τεχνικά μέρη του αυτοκινήτου. Και κατά την άποψή μου λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να ασχοληθεί με αυτά τα γενικότερα δεδομένα. Αυτά τα γενικότερα ζητήματα πρόσβαση στα τεχνικά δεδομένα. Με ανησυχεί το γεγονό λοιπόν ότι έχουμε μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση, ότι συζητούμε το ένα ζήτημα μετά το άλλο. Και καταλαβαίνω λοιπόν το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τα στις υπηρεσίες τις εμπορικές, αλλά πιστεύω ότι η δικιά μας η προσέγγιση, η δικιά μας η αρμοδιότητα εδώ είναι να δημιουργήσουμε ένα ε, δημόσιο σύστημα ανώνυμο υψηλής ποιότητας με βάση την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποιες αναφορές στις αιτιολογικές σκέψεις, αλλά όχι στα άρθρα του κανονισμού κατά την απόψή μου, γιατί τα θέματα αυτά εκφεύγουν τελείως του πεδίου εφαρμογής του. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Για να πάρουμε το λόγο με τη σειρά των παρεμβάσεων και για να απαντήσω στα τελευταία σχόλια που κάνατε κατευθείαν. Η απάντησή μου είναι η εξή. Τρία διαφορετικά στοιχεία έχω να παρουσιάσω. Θα είμαι σύντομο. Η ιστορία αυτή ασφαλώς έχει και μία ιστορία. Ξεκίνησε με την ιδέα του πειραματικού το 2006 στην ομάδα 29 αναφέρθηκε αυτή η ανησυχία σε ένα έγγραφο εργασία το οποίο πλέον αναφέρεται σε μία από τις αιτιολογικές σκέψεις. Αυτή η ανησυχία λοιπόν οδήγησε σε κάποιες αντιδράσεις, σε κάποιες βελτιώσεις. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστό να λέμε ότι η πληροφορία που ενέχεται στο 112 το e-call ανωνυμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ισχύει η οδηγία για την προστασία δεδομένων. Μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά σχετίζεται με την ε, συμπεριφορά του οχήματο. Δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο οδηγός με σιγουριά. Ξέρουμε όμως ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ο συνήθις οδηγός. Και σε έναν κόσμο με τόσο δεδομένα η ανάλυση των ε, συστημάτων ε, ε, οδήγησης κυκλοφορίας. Όσο πιο πολλά πληροφορίε έχουμε, τόσο πιο πολύ είναι, πιο σωστή είναι η υπόθεση. Τώρα να περάσουμε σε ένα υποχρεωτικό σύστημα e-call, το οποίο θα αποτελεί στην πλατφόρμα για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Ναι, λοιπόν, αυτό ισχύει και γι' αυτό γίνονται αυτές οι αναφορές. Καταλαβαίνω λοιπόν το επιχείρημα ότι η πρόταση επικεντρώνεται στο υποχρεωτικό δημόσιο e-call, αλλά στις συντολογικές σκέψεις έχουμε ήδη περάσει αυτό το επίπεδο, αυτή τη γραμμή. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αναφέρθηκε επαναλημμένα ότι το θέμα αυτό είναι μόνο για να δοθούν ισχυρά και χειρά μηνύματα στις συντολογικές σκέψεις 6, 7, 8, 9. Αυτό αναφέρεται στην πραγματικότητα αυτή και ήδη προβλέπει μια υποχρέωση για να δίδονται τέτοιες πληροφορίες σε αυτή την κοινή δημόσια βάση την υποχρεωτική βάση. Αυτό για το 3-1. Και γίνεται αυτό και στο διατακτικό. Με το ίδιο λοιπόν, με την ίδια λοιπόν σκέψη και την ίδια αιτιολογία, αν υπάρξει αυτή η εξέλιξη, θα, αποτελεί, θα αποτελέσει αυτό το βασικό κατόφλι σε ένα περιβάλλον, και θα χρησιμοποιήσω μια δυνατή λέξη, περιβάλλον επιτηρήσεις Το κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τέτοια θέματα τώρα. Δεν λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία υπερβολική αντίδραση, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα πιο βασικά στοιχεία προκειμένου να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση. Και αυτό λοιπόν χρησιμοποίησα ε, αυτό το επιχείρημα σε ό,τι αφορά το χάρτη, χάρτα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 16 της ε, συνθήκης. Και μας δίνει και η καθοδήγησή μας αν λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το e-call δεν θα οδηγήσει σε διαρκή παρακολούθηση, θα μπορούσαμε εκ παραλλήλου να πούμε ότι αυτό θα αποτελέσει ελάχιστο πρότυπο για το ιδιωτικό e-call, ότι δεν θα πρέπει να ωφελούνται λοιπόν από την διευκόλυνση αυτή. Αν γίνει τέτοια αναφορά στην ανάγκη να διασφαλιστεί εθελούσια συμμετοχή όπως αναφέρεται στην τροπολογία 6, το κείμενο αυτό θα είναι πάρα πολύ απλό και δεν θα συνεχιστεί εκτός και αν συμπεριληφθεί στις α, όρους έγκρισης, ότι θα πρέπει να υπάρχει η τεχνολογία για να συμβούν αυτά. Ιδάλλως δεν πρόκειται απλά να συμβούν. Αυτό λοιπόν θα σας απευθύνω ως έκκληση. δεν θέλω να ξεφύγουμε σε κάτι που δεν θα είναι ρυθμισμένο. Όχι, υπάρχει μια γενική οδηγία, γενική όρη, θα ισχύουν στους operators. Τα προβλήματα λοιπόν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν ενεργά. Εκ των προτέρων, ιδάλλως θα προκληθούν όλο και πιο πολλές τριβές, οι οποίες θα αποβούν προς ε, εις βάρος των χρηστών, θα βλάψουν και τελικά το σύστημα 112 είναι ένα καλό παράδειγμα δημόσιων υποδομών που δημιουργούνται για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον α, υπηρεσιών που θα είναι αποδεκτές. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει στο άρθρο 6, 6 σε κάποιες αντιλογικές σκέψεις και προφανώς ε, θα δώσει ο, ο νομοθέτης κάποια καθοδήγηση και θα υπάρξει κάποια ρύθμιση προφανώς. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε δύο πράγματα. Να πούμε ότι, α, κοιτάξτε, είναι εκτός του πλαισίου και μετά να εισαγάγουμε διατάξεις οι οποίες οι ίδιες να ξεφεύγουν από το πλαίσιο. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν μια υποδομή αποδεκτή και αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα, στην παρούσα χρονική συγκυρία και θα δούμε τέτοια παραδείγματα πολλά στο μέλλον, όπου η τεχνολογία θα έρχεται έτσι σε άλλη επικάλυψη με το ρυθμιστικό περιβάλλον και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά θα γίνουν με τον σωστό τρόπο. Και μπορούν να γίνουν με σωστό τρόπο, με έναν τρόπο που να μην προκαλέσει κατακαιρματισμό της αγοράς. Και αυτό θα πρέπει να απασχολεί την αγορά σας. Αν δεν το διευκρινίσετε αυτό, θα δημιουργηθεί, θα γίνει αυτό με κατακαιρματισμένο τρόπο και θα προκαλέσει ενοχλήσεις. Γιατί λοιπόν να μην γίνει αυτό με τόσο σωστό τρόπο για την ιστορική αγορά, για την προστασία των δεδομένων, για τη καλή λειτουργία της αγοράς και των καταναλωτών, προστασία των καταναλωτών. Άρα λοιπόν, τι να σας πω, ακολουθήστε τη ροή της τεχνολογίας. Λυπάμαι, Πρόεδρε. Ναι, δεν ναι, ναι, ξέρω, λέει ο Πρόεδρος, απλά ελέγχω την ισχύ των επιχειρημάτων σας. Κοιτάξτε, δεν είναι κόλπα αυτά. Να ακούσουμε και τους άλλους δύο μιλητές. Ο κύριος Όμπερμαϊερ θέλει να κάνει ερωτήσεις. Να ακούσουμε όμως πρώτα τον κύριο Ρουκ και την κυρία Διάννη. Και μετά θα κάνουμε ένα δεύτερο γύρο. Σχετικά με τις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν για την κυρία Σενάλοβα. Τα κράτη-μέλη τα οποία είναι εκτός της οικογένειας Χέρο είναι δύο ομάδες βασικά, χονδρικά. Καταρχάς οι χώρες οι οποίες δεν υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός συστήματος πανευρωπαϊκού για οικονομικούς κυριολόγους και αυτό περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει και μια άλλη ομάδα η οποία στηρίζει ένα πανευρωπαϊκό οίκομα αλλά δεν έχουν καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και χρειάζονται βοήθεια γιατί μιλάμε για ένα πολύ εξειδικευμένο σύστημα το οποίο κάνει μια πολύ συγκεκριμένη, φέρει πέρας μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε ε, με ε, χώρες μέλη οι οποίες στα πλαίσια της διατύπωσης των συγκεκριμένων τεχνητών απαιτήσεων και ρυθμίσεων έχουν ήδη πάρει μέρος στην προετοιμασία του συστήματος. Το πρόγραμμα Hero υπάρχει, υπάρχει για πολύ συγκεκριμένους λόγους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη βοήθεια. Για το αν θα είμαστε έτοιμοι τώρα το 2015. Υπάρχουν τρία βασικά εδώ στοιχεία. Καταρχάς, οι κατασκευαστές σε αυτοκινητοβιομηχανίες εμπλέκονται στα πλαίσια του e από το 1998. Δεν είναι κάτι νέο για αυτούς, τα περισσότερα οχήματα κατασκευάζονται σε παγκόσμια κλίμακα και αυτό περιλαμβάνει και τη Ρωσία. Και το ρωσικό σύστημα, το οποίο είναι σχεδόν ταυτόσιμο με το δικό μας, θα αναπτυχθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Τα οχήματα δηλαδή με e-call θα αρχίσουν έτσι και αλλιώς πριν από μας να κυκλοφορούν στη Ρωσία. Τα στοιχεία τα οποία δίνουν είναι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη πράγματι και απαιτούν περισσότερο χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά εμπλέκονται στην προετοιμασία του e-call εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα για τα ασύρματα δίκτυα κινητό, κινητής τηλεφωνίας. Η κατάσταση ποικίλει από χώρα σε χώρα. Το βασικό στοιχείο είναι ότι πρέπει να, να επιτρέπουν στο σύστημα να κρίνει όταν μία α, κλίση φωνητική περιλαμβάνει εσωτερικά δεδομένα. Τα κινητά δίκτυα τα PSAAP λοιπόν θα πρέπει να επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν και να επιτρέψουν την αναβάθμιση. Αυτά για τις ερωτήσεις της Σενάλοβα. Ε, θέσατε επίσης και το θέμα του κόστους της εκκίνησης της διαδικασίας. Νομίζω ότι εδώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική, ε, ε, ένας διαφορετικός υπολογισμός του κόστους. Το αρχικό κόστος για το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ. Το πραγματικό κόστος είναι 300.000 ευρώ. Εγώ είμαι σε στενή επαφή, σε εβδομαδία βάση με τους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρέχουμε σύνδρομη όπου μπορούμε και παρακολουθούν από πάρα πολύ κοντά το τι συμβαίνει με το πρόγραμμα Hero. Τώρα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πολλοί κατασκευαστές οχημάτων ε, συζητούν τη χρήση ενός οδηγικού συστήματος αν θέλετε. Τμήμα της τηλεματικής τους πλατφόρμας θα περιλαμβάνει το σύστημα e-call με τον κλίση 112 σαν ξεχωριστό κομμάτι το κομμάτι το οποίο αφορά τις εμπορικές ε, χρήσεις και εφαρμογές δεν χρησιμοποιεί την ενυπνώση SIM. Πρόκειται για μια επιμέρους εμπορική συμφωνία. Όμως, αυτή είναι η τάση θα έλεγα για κάποιους από τους κατασκευαστές ε, οχημάτων ιδιαίτερα ε, σε σχέση με τα ακριβά μοντέλα τους. Μία πλατφόρμα, δύο εφαρμογές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να επιβεβαιώσω ότι από το δικό μας παρατηρητήριο σε ό,τι έχει σχέση με το έγνος και από, τη, από το 2009 που υπάρχουν κάποιοι δέκτες συμβατοί με το έγνωσο δεν υπάρχουν προβλήματα με τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Για το Γαλιλαίο. Αυτό το οποίο απαιτείται στην πρόταση κανονισμού για την έγκριση τύπου είναι φυσικά η συμβατότητα. Συμβατότητα λοιπόν με τον Γαλιλαίο μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια ε, των ε, ήδη υπαρχουσών ε, συστημάτων ελέγχου ανάμεσα σε διαφορετικές μονάδες. Και ήδη υπάρχουν προϊόντα στην αγορά τα οποία διαφημίζονται ότι είναι συμβατά με τον Γαλιλαίο και υπάρχουν και άλλα πρότυπα τα οποία προσπαθούν να γίνουν συμβατά με το πρότυπο Γαλιλαίο. Συνεπώς λοιπόν δεν θα υπάρξει πρόβλημα για μας σε σχέση με αυτά τα συστήματα εγκαίρως να κυκλοφορήσουν εγκαίρως. Πρέπει όμως οι διαδικασίες να επιταχυνθούν. Well, I think um, we've had a very um, good Ωραία. Ήταν νομίζω όμορφη αυτή η ενταλλαγή απόψε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Μήπως η Επιτροπή. Όχι. Μάλλον καλύψαμε το θέμα. Κυρία Σεναλόβα. Εσείς αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία. Μήπως θέλετε να κλείσετε με ένα συμπέρασμα. Νομίζω συλλέξαμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να λάβουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Ε, στην πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, ήταν πολύ χρήσιμη για όλους. για όλους εκείνους που ασχολούνται με το θέμα αυτό εδώ και χρόνια και με χαρά διαπίστωσα ότι ε, έχει σημειωθεί πρόοδος. Ε, εκτιμώ τις παρατηρήσεις ε, του ελεγκτή προσωπικών δεδομένων. Έχουμε λάβει πάνω από 100 τροπολογίες, 37 έχω υποβάλει ως εισηγήτρια. Οι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες αναφέρονται κυρίως ε, στα σχόλια, στις παρατηρήσεις ε, ε, του επόπτη προσωπικών δεδομένων του κ. Χάστινγκς. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς με την αξία του ε, δημόσιου συστήματος e-call για κλήσεις έκτακτης ανάγκης 112. Υπάρχει μια γενική συμφωνία λοιπόν με τις θέσεις σας. Το... Ε, στην τροπολογία θα τη συζητήσω με τους ε, σκιώδεις ηγητές μαζί και με τις δικές σας παρατηρήσεις την επόμενη εβδομάδα. Αναμένουμε επίσης και τις τροπολογίες από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευελπιστώ λοιπόν ότι θα βρούμε μια λύση. ώστε η τελική έκθεση που θα υποβάλουμε να αντανακλά όλες αυτές τις απόψεις που εκφράστηκαν. Ανάμεσα σε αυτές και τις δικές σας παρατηρήσεις. Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη μήνυα ακρόαση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ την πλευρά μας για την συμμετοχή. και ολοκληρώσαμε τις εργασίες της ε, Επιτροπής μας. Για σήμερα η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 10, 16 και 17 Δεκεμβρίου. Δευτέρα και Τρίτη. Τη Δευτέρα από τις 3 μέχρι τις 6.30 και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου θα έχουμε την ψηφοφορία το πρωί από τις 9 μέχρι τις 12.30 και άλλη μια σύνοδο από τις 3 μέχρι τις 6.30. Και αν θυμάμαι καλά, την ψηφοφορία για τη δικιά σας πρώτη κυρία Συναλαβά θα την κάνουμε τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Thank you, Olga. I think everybody knew your timetable anyway. I just have it here. Yeah. Yeah. Yeah.